Θα ξεκινήσω ζητώντας να εγκρίνετε την ημερήσια διάταξη. Δεν ζητήθησαν αλλαγές για την ημερήσια διάταξη. Να σας πω ότι θα προβώ σε ανακοινώσει της Προέδρου αργότερα. Έχουμε ελάχιστο χρόνο για το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Τι ανακοινώσει θα τι αφήσουμε για αργότερα. Ξεκινάμε τη συνεδρίαση. Με το, με το σημείο το, που έχουμε να συζητήσουμε και έχουμε τον εκπρόσωπο τη Ασκφώση για στρατηγικά θέματα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το δημοψήφισμα ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Τζόναθαν Φολ. Πριν ξεκινήσουμε, να πω ότι θεωρείται η μερίσια διάταξη με αυτή τη μικρή αλλαγή που σας ανέφερα ως εγκεκριμένη, ε, διότι δεν ζητήθηκε κάτι διαφορετικό. Το τρίτο και τέταρτο σημείο θα συζητηθούν αργότερα έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 28 Σεπτεμβρίου και 22 Οκτωβρίου έχουν διατεθεί ως συνήθως και θεωρούνται εγκεκριμένα αν δεν προβληθεί αντίρρηση μέχρι το τέλος συνεδριάσεως. Να σας ενημερώσω ότι ως ήθιστε η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο και πάμε στο σημείο 6 της ημερησίας διατάξεως οι διαπραγματεύσει με το Ηνωμένο Βασίλειο, συνταγματικέ σχέσει του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σοβαρότατο ο τίτλο. Θα ζητήσω τον Τζόναθαν Φαουλ που είναι επικεφαλή τη Task Force για στρατηγικά θέματα που σχετίζονται με το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, να πάρει το λόγο και μετά θα ακούσουμε ερωτήσει, απαντήσει και σχόλια. Τζόναθαν, ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή χρονιά σε όλους. Όπως γνωρίζετε, ο Βρετανός Πρωθυπουργό σε μια επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Τούσκ, ανέφερε τέσσερις κατηγορίες θεμάτων, τέσσερα καλάθια που τα αποκαλεί, με θέματα που θέλει να συζητηθούν. Η επιστολή απεστάλλει τη 10η Νοεμβρίου, έκτοτε διεξήχθησαν εντατικές συζητήσεις, κάποιες άτυπες, κάποιες επίσημες και στις Βρυξέλλες αλλά οι υπουργοί, διπλωμάτες ε, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ταξίδεψαν στην Ευρώπη και συνομίλησαν με τους ε, ομολόγους τους. Διεξήχθη Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον μήνα Δεκέμβριο. Θα υπάρξει και άλλο στις 18 και 19 Φεβρουαρίου και το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενδεχομένως θα είναι εκείνο στο οποίο θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις από του θέματος. Σίγουρα το θέμα αυτό είναι στην ημερήσια διάταξη, διεξάγονται εντατικότατες συζητήσεις τώρα και μέχρι τότε, ούτω ώστε να βρεθεί καλύτερη δυνατή λύση. Θα γνωρίζετε ότι ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει θεσπιστεί νομοθεσία για τη διοργάνωση του δημοσιφίσματος, διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες στο νέο αυτό νομοσχέδιο και θα πρέπει να διεξαχθεί μέχρι τέλος του 2017 το δημοψήφισμα. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, μπορεί να διεξαχθεί και νωρίτερα. Αυτό θα το αποφασίσουν οι Βρετανοί. Όμως θα παρακολουθείτε στα μέσα ενημέρωση τα της η οποία ξεκινά πραγματικά και πιο επίσημα θα ξεκινήσει από τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις και θα καθοριστεί επισήμως η ημερομηνία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απλούστατη, θέλουμε στην υποκοδομητική. συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους της Γραμματείας του Συμβουλίου, επιδιώκουμε να σας ενημερώνουμε στο βαθμό του δυνατού ούτως ώστε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να συνεργάζονται και να προβάλλουν και αυτή την εικόνα και παίζουμε και ρόλο στην εξέβρεση λύσεων στα θυγέντα προβλήματα συνδεόμενοι με τα άλλα 27 κάτι μέλη ούτως ώστε να αντικατοπτρίζονται και τα δικά του συμφέροντα ω αρμόζει στα αποτελέσματα που θα προκύψουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εκεί θα ληφθεί απόφαση με συνένεση. Έχουμε κρίσιμη συνεδρίαση που επίκειται. Θα γίνει σύντομα. Αν δείτε τι έγινε με αντίστροφη πορεία από την ημερομηνία που θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα χρειαστεί έγγραφα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, άρα αρχές Φεβρουαρίου, κινούμενοι πάντα αντίστροφοι χρονικά, θα πρέπει να συνταχθούν τα έγγραφα και το όλο θέμα τότε θα συζητηθεί δημοσία σε όλα τα κράτη-μέλη. Έτσι έχουν τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να βοηθήσει ως θεματοφύλαξη των συνθήκων, θέλει να εξασφαλίσει ότι το νομικό σύστημα της ενός θα διατηρηθεί ως έχει για να προδικάσω την ερώτηση που προβλέπω τα τεθεί. Τι μορφή θα έχει η απόφαση, η διευθέτηση, η λύση. Η μορφή θα ακολουθεί στο περιεχόμενο βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει φάσμα δυνατοτήτων. Πικίλη; από απλές δηλώσεις του Συμβουλίου, διακηρύξεις, ίσως να γίνουν παραπομπές σε νομοθετική δραστηριότητα, κάτι που αφορά το κοινοβούλιο είναι το χρόνο, ίσως και όχι, εξαρτάται από τα δέοντα. Δεν θα σας αποκρύψω ότι πρέπει να συζητηθεί και το ενδεχόμενο τροποποίησος της συνθήκης, των συνθήκων. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να πηρηθούν τα θέματα εντός των παρουσών συνθήκων ή δυνατών. Όλα αυτά θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και οι ελπίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι αυτό το Συμβούλιο θα αποδεικτεί ότι είναι και το αποφασιστικό. Ευχαριστώ πολύ. Ήδη έχω 11 συναδέλφους που επιθυμάνε να λάβουν το λόγο. Εστέλα Κονική παρακαλώ, διότι έχουμε μόνο μέχρι τις 11 χρόνο για συζήτηση. Και θέλω να μιλήσουν όλοι. Ο Πολ Ρέιντζολ, ο είναι εδώ. George Σέπλιν. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, καλώς ήρθατε κύριε Φόλ. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Μία ερώτηση έχω. Ε, πιο σημαντική θεωρώ εγώ. Η διασφάλιση των τεσσάρων ελευθεριών. Ελπίζω ότι η δουλειά που κάνετε είναι να αναζητείτε λύσεις. Ε, αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, δηλαδή να αντιληφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο ότι αυτές είναι απαραβίαστες. Εντάξει, κάποιες μικρολεπτομέρειες, αλλά δεν υπάρχει τρόπος, ε, δεν είναι δυνατόν δηλαδή, να παραβιαστούν τέσσερις ελευθερίες. Ναι ή όχι. Ναι, συμφωνώ. Μάλιστα, Μερσέντες Βρέσο. Ευχαριστώ. με ικανοποίηση λαμβάνω υπόψη την πρώτη απάντηση επί του θέματος των τεσσάρων ελευθεριών. Από ό,τι κατάλαβα, από αυτά που είπατε εντάχει, και η Βρετανική κυβέρνηση θα προτιμούσε μια δήλωση, μια διακήρυξη που ενδεχομένω θα περιείχε παραπομπή σε νομοθετικές τροποποίησεις που θα παραστούν αναγκές. Καλύτερο αυτό παρά τροποποίηση των συνθήκων. Διότι είναι σαφές ότι το χρονικό ζήτημα είναι σημαντικότατο. Όμως, κατά την άποψή σας, αρκεί πολιτική συμφωνία με μια δήλωση που είναι το πρώτο ενδεχόμενο. και εκεί θα μπορούσε να αποστεθεί και ένα παράρτημα με ανάληψη δέσμευσης για μια διαδικασία για κάποιες τροποποίησεις. Για να καταλάβω το θέτω το ερώτημα. Διαφορετικά αυτό θα σήμαινε ότι αν χρειάζεται τροποποίηση των συνθηκών αυτό θα μπορεί να συμβεί μόνο μετά το δημοψήφισμα με καμία εγγύηση για τα δύο μέρη. Ούτε για την υπόλοιπη Ευρώπη Η τοπή των συνθηκών μπορεί να τροποποιήσει το αποτέλεσμα χωρί καμία εγγύηση όμω για του Άγγλου που δεν θα γνωρίζουν αν η τροποποίηση των συνθηκών τελικά θα λάβει χώρα πραγματικά ή όχι. Άρα υπάρχει τάση να βρεθεί λύση εντός των συνθηκών. Με τον συνάδελφο Μπροκ ετοιμάζω μια έκθεση. Η έκθεση δείχνει ότι πολλά πράγματα μπορούν να γίνονται των ηθικών. Συνεπώς αυτό θα μπορούσε να είναι πιο λογική η λύση για όλους. Θα μπορούσε να επιτρέψει την εξέβρεση λύσεων πάντα στα πλαίσια της πράσπης των τεσσάρων ελευθεριών και λύσεις οι οποίες θα είναι καλές για όλους. Thank you. Uh, if... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν κατάλαβα καλά την αρχή της ερώτησης, με ρωτήσετε τι προτιμάει η Βρετανική κυβέρνηση. Ε, δεν το ξέρω αυτό. Δεν είναι η δικιά μου δουλειά. Ξέρουμε ότι ο Πρωθυπουργό είπε ότι θέλει νομικά δεσμευτικές και ε, μη αναστρέψιμες λύσεις. Αν δούμε λοιπόν τα διάφορα πιθανά μέσα που κυμαίνονται από δηλώσεις, ε, αποφάσεις εντός του υφιστάμενου πλαισίου ε, μέχρι νομοθεσία, μέχρι και αλλαγή της συνθήκης τότε προφανώς υπάρχουν ζητήματα χρόνου και τελικά η επιλογή θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνουμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα, πολλές ε, απαντήσεις θα έλεγα στις βρετανικές ανησυχίες εντός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και αυτό μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα. Μπορεί να υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν την νομοθεσία που χρειάζονται βεβαίω κάποιο χρόνο όπως ξέρουμε και οπωσδήποτε το ίδιο ισχύει και για την αλλαγή της συνθήκης. Και εδώ εντός του θεσμικού πλαισίου της Ένωσης και στα κράτη-μέλη σύμφωνα με το σύνταγμά τους. Τα πάντα λοιπόν θα εξαρτηθούν από το τι θα γίνει και δεν μπορώ σήμερα να σας πω κάτι οριστικό γιατί δεν ξέρω ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μόνο τότε θα αποφασιστεί το πώς θα εφαρμοστούν νομικό ζήτημα οπωσδήποτε, αλλά με σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε, γιατί έχει ξαναγίνει, είναι πως μία απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ήδη μια συμφωνία κάποια αποτελέσματα και η αφετηρία είναι ελπίζω ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα καταλήξουν σε συμφωνία επί κάποιων πραγμάτων που μετά θα πρέπει να εφαρμοστούν αναλόγως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαίτερ Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά έχουμε επίγνωση ότι δεν μπορείτε ακόμη να μας δώσετε συγκεκριμένες πληροφορίες παρά μόνο περισσότερες γενικές παρατηρήσεις και φυσικά την διαφύλαξη των τεσσάρων ελευθεριών, όπως είπε και ο κύριο Σέπφλινγκ. Και σίγουρα υπάρχει ένα τμήμα που αφορά τις διατάξεις, τους κανονισμούς, αυτό το επεξεργάζει το Συμβούλιο, αλλά έχουμε και ε, στοιχεία, δεδομένα. Το φλέγον ζήτημα, το καθόντε ζήτημα των κοινωνικών επιδομάτων, εργασιακών επιδομάτων των ξένων υπηκών που εργάζονται στο Ηνωμένο, Βασίλ... στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί υπάρχουν στοιχεία πόσοι ξένοι υπήκοοι Ευρωπαίοι βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, πώς εργάζονται, πώς είναι δικαιούχοι κοινωνικών ε, επιδομάτων. Για να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα και να ξέρουμε περί τίνο πράγματο μιλάμε, περί τίνο πρόκειται. Γιατί επιμένει πολύ σε αυτό το θέμα των κοινωνικών επιδομάτων ε, το Ηνωμένο Βασίλειο. Και το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο και για το Ηνωμένο Βασίλειο και για τους ε, Ευρωπαίους πολίτες γενικά. Γιατί ζητά κατάργηση ο Κάμερον για τους ξένους υπηκόους, αλλά θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα, αλλά από στοιχεία συγκεκριμένα τίποτα. Έχετε κάποια τέτοια στοιχεία στη διάθεσή σας για να ξέρουμε γιατί ακριβώς μιλάμε. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν ε, πολλά στοιχεία για τον αριθμό των υπηκών άλλων κρατών μελών που δουλεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντιστρόφως βεβαίως για τους Βρετανούς σε άλλα κράτη-μέλη. Και ευχαρίστως να σας δώσω αυτά τα δεδομένα. Ο αντίκτυπος σε αυτούς τους ανθρώπους βεβαίως εξαρτάται από το τι θα αποφασιστεί και πρέπει να το σκεφτούμε προσεκτικά οπωσδήποτε έδωσα μια σύντομη απάντηση πριν στο ερώτημα του κυρίου Σεφίν. οι θεμελιώδης ελευθερίες είναι θεμελιώδεις και εμείς αλλά και οι Βρετανοί νομίζω θα έλεγαν πως α, παίρνουν πολύ σοβαρά αυτά οι θεμελιώδεις ελευθερίες ε, δεν είναι ανεφόρον η συνθήκη και η παραγωγός νομοθεσία ορίζουν κάποιους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους εργαζόμενοι και αγαθά και κεφάλαια και υπηρεσίες ε, έχουν αυτές τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες. Εξετάζουμε λοιπόν πολύ σοβαρά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και το ζήτημα είναι το οποίο θα κρίνει δηλαδή τη μορφή τυχών αλλαγών το εάν υπάρχει επαρκής ευελιξία στο υφιστάμενο πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά τηρώντας ε, προφανώς ε, τις ε, βασικές αρχές τις τέσσερις βασικές ελευθερίες που πρέπει να παραμείνουν άθικτες. Ευχαριστώ κύριος Μασέρσμιτ. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να εστιαστώ σε ένα από τα πράγματα που αναφέρατε στην αρχή στον ρόλο των κρατών μελών. Το Ηνωμένο Βασίλειο είπε πως θέλει να αλλάξει την διαδικασία της ε, κίτρινης ε, και πορτοκαλί κάρτας σε κόκκινη κάρτα. Μπορεί να γίνει αυτό χωρίς αλλαγή της ε, συνθήκης. Τι σκέψη έχετε κάνει για την περαιτέρω εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων στην νομοθετική διαδικασία. Ναι. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για το θέμα αυτό και γνωρίζουμε ότι πολλοί μηχανισμοί θεσπίστηκαν ε, επί σειρά ετών ε, προκειμένου να μειχθούν και τα εθνικά κοινοβούλια στη διαδικασία λήψη αποφάσεων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς βέβαια να παρεμποδιστεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου που είναι οι συνομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολλά θέματα συζητήθηκαν και προτάσει για το πώς θα βελτιωθεί το τρέχον σύστημα προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων. Τώρα, τι μηχανισμός θα χρησιμοποιηθεί για να εφαρμοστεί μια τέτοια συμφωνία θα εξαρτηθεί από την ουσία της συμφωνίας αυτής, από το περιεχόμενό της. Και προς το παρόν δεν έχουμε τέτοια συμφωνία. Δεν κάνω το δύσκολο, θέλω να είμαι ιδιότροπος, αλλά πραγματικά δεν ε, γνωρίζω αυτό το θέμα ακόμη. Θα εξαρτηθεί από το σε τι βαθμό θα τροποποιηθούν οι ισχύοντες κανόνες. Και πολλές προτάσεις υπάρχουν για τις σχέσεις μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Όταν επιτευχθεί συμφωνία, για το τι μέλη τότε θα πρέπει να δούμε και πώς ε, θα εφαρμόσουμε τη σχετική συμφωνία. Ο Χέλμοντ Σόλτς. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ μια ερώτηση για το θέμα αυτό του δευτερογενούς δικαίου, του παραγόγου δικαίου. Μιλήσατε για τις τέσσερις ελευθερίες, αλλά στην επιστολή Κάμερον τίθεται πράγματι το ζήτημα της ελεύθερης ε, διακίνησης. Και πράγματι εδώ πέρα ίσως απαιτηθεί μια αλλαγή της ε, συνθήκης. θα απαιτείται σε αυτή την περίπτωση μία δεβαίωση των 27 υπολείπων κρατών μελών ε, απέναντι στην Βρετανία, η οποία μάλλον δεν μπορεί να έρθει πριν από το δημοψήφισμα. Και τέλος, το θέμα είναι πάρα πολύ ε, επίκαιρο γιατί υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ε, πολιτικής που ακολουθείται Και μην ξεχνάμε, η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει υπογράψει τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι νομική βάση για πολλούς ε, πολίτες και ενισχύουν αυτή την εμπιστοσύνη. Τι, πώς το βλέπετε το δημοψήφισμα, το δημοψήφισμα σε σχέση με την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Um, the of... Ευχαριστώ. Η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, δεν ανέκυψε στη συζήτηση, ούτε αναφέρεται στην επιστολή του Πρωθυπουργού. Θα ήθελα να επαναλάβω πως δεν είμαι βέβαιος ότι η ικανοποίηση των ε, ε, ετοιμάτων των νησιών του Βρετανού Πρωθυπουργού ε, ότι δεν απαιτεί συνταγματικέ αλλαγέ, αλλαγέ τη συνθήκη, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια τέτοια διαδικασία χρονοβόρα, απαιτεί κύρωση από τα κράτη-μέλη. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο βασικό λόγο ε, τη ανάλυση τη ερώτηση. Το θέμα είναι τι θα συμφωνηθεί, ποιο θα είναι το περιεχόμενο τη συμφωνία και κατόπιν πώ θα εφαρμόσει τη συμφωνία αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει ένα ευρύ φάσμα του πιθανού περιεχομένου και για πολλά θέματα, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να βρεθεί λύση χωρίς παραβίαση της υφιστάμενης συνθήκης ή των υφιστάμενων συνθήκων και χωρίς να απαιτείται και τροποποίηση αναθεώρηση των συνθήκων. Αλλά θα δούμε, γιατί σε τελική ανάλυση αναπόκειται στους αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων να αποφασίσουν τι πρέπει να γίνει και μετά θα αποφασίσουμε οι υπόλοιποι πώς θα το εφαρμόσουμε τον καλύτερο τρόπο. Ο κύριος Καστάλντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι απλή και περίπλοκη η ερώτησή μου ταυτόχρονα όσον αφορά την παρούσα κατάσταση, το πολιτικό πλαίσιο σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Διερωτώ με μήπω υπάρχει κάποιο κίνδυνο Η απάντηση, αν καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα και συμφωνία και πρέπει να εφαρμοστεί. Και μήπω έχουμε αποτέλεσμα ντόμινο, δηλαδή και άλλα κράτη ευρωπαϊκά τελικά να θελήσουν να προωθήσουν παρόμοια αιτήματα. Να ζητήσουν να εξαιρεθούν από κάποιες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ή να αναδιαπραγματευτούν το, το καθεστώς υπό το στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνατε κάποια ανάλυση. Έχετε προετοιμάσει στατηγική για τέτοια ενδεχόμενα. Τι αντιδράσεις μπορεί να προβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν από άλλες χώρες, Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία, από άλλη χώρα καταφτάσουν παρόμοια αιτήματα. Αυτοεξαιρέσεων, opt-out από τις συνθήκες ή διαπραγματεύσεις νομοθετικού περιεχομένου για να δημιουργηθούν ιδιαίτερα καθεστώτα για κάθε χώρα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, υπάρχει μια θεμελιώδης επιλογή πρέπει να γίνει. Πρέπει να δούμε αν οι αλλαγές, οι δηλώσεις που θα γίνουν σαν απάντηση στις ανησυχίες του Βρετανού Πρωθυπουργού αφορούν αποκλειστικά το Ηνωμένο Βασίλειο ή αν θα είναι γενικές αντιδράσεις. Εν τη αυτή ο οδήποτε κράτος μέλος μπορεί να ωφεληθεί αν το επιθυμεί. Αυτό αφορά τα κράτη-μέλη. Ε, πολλά από τα ζητήματα που θίγει ο Πρωθυπουργό στην επιστολή του θα οδηγήσουν σε δηλώσεις και αναλήψει υποχρεώσεων ενδεχομένως που ίσως να είναι διαθέσιμα ως και σε αλλα κάτι κράτη-μέλη. Αν δημοκρατικά τα άλλα κράτη αποφασίσουν να ακολουθήσουν παρόμοια πορεία, αυτό αφορά τα κράτη. Για να απαντήσω στην άλλη ερώτησή σας. Αν άλλα κράτη-μέλη υποβάλλουν ε, αιτήματα και θέματα, τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ακούσει με σεβασμό τα κράτη-μέλη όταν θα εκφράσουν ανησυχίες. Ε, θα εφαρμόσουν το κράτος δικαίου, τις συνθήκες ως ισχύουν, την ισχύουσα νομοθεσία. Και αυτή είναι εξαιρετική περίσταση. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ένα κάτος μέλος αποφάσισε να διεξαγάγει δημοψήφισμα περί παραμονής ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και εμείς θα αντιδρούμε σε αυτό το γεγονός. Σας ευχαριστώ, David McAllister. Ευχαριστώ. Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο δύσκολες ήταν μέχρι στιγμής οι διαπραγματεύσεις στην πράξη. Και δεύτερη ερώτηση. Ε, ε εντάξει, δεν θέλω τώρα να κάνω το πράκτορα πολυφυλαχιών, αλλά πόσο πιθανό είναι να έχουμε μια τέτοια συμφωνία το Φεβρουάριο. Δεν θέλω να είμαι εγώ ο ένοχος ή ο υπεύθυνο για τα, τα στοιχήματα που βάζετε ή τις αλλά υπάρχει, υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες για λήψη απόφασης το Φεβρουάριο. Και φαίνεται η βούληση των αρχηγών να επιλύσουν το θέμα, αλλά φυσικά χρειάζεται ο χρόνος για να γίνει κάτι τέτοιο. Και μέχρι το Φεβράριο λίγε εβδομάδε μόνο μα έχουν απομείνει και υπάρχουν ακόμη ακαθόδη ζητήματα που παρέμειναν εκκρεμή. Και εγώ δεν συνηθίζω να στοιχηματίζω, ούτε πρόκειται να βάλω στοίχημα και δεν θα σας εθένα ούτε και εσάς να στοιχηματίσετε σε αυτό. Πάντως, από ό,τι βλέπω, η πολιτική βούληση για την επίλυση του θέματος ε, είναι αρκετά σημαντική. Αλλά θα δούμε. Τώρα, για την πρώτη ερώτηση που είναι συναφής με τη δεύτερη, ήταν δύσκολες οι πραγματεύσεις ε, και από πολιτική και από νομική άποψη. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρχαν δυσκολίες, αλλά και στις υπόλοιπες 27 ε, χώρες μέλη. Και υπάρχουν δυσκολίες και νομικές ως προς το νομικό σύστημα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να εφαρμόσει. Το θέμα είναι ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και των υπολείπων, πώς λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις η εσωτερική αγορά, το θέμα της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ε, εργάζονται ή πώς τους μεταχειρίζονται οι χώρες μέλη τους εργαζόμενους ε, στην επικρατειά τους και πολλές απόψεις ε, διατυπώθηκαν για τα θέματα αυτά. Σίγουρα λοιπόν δεν ήταν καθόλου εύκολες οι διαπραγματεύσεις, ούτε έχουμε φτάσει σε κάποιο συμπέρασμα. Πάντως το ενθαρρυντικό είναι η ισχυρή επιθυμία και βούληση για επίτευξη λύσης και μάλιστα χωρίς να θυσιάσουμε όλα τα κεκτημένα, όλα τα καλά και τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω μία αθώα ερώτηση για την ατμόσφαιρα που κρατεί στις Από μία πρώτη ματιά, η Ένωση αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα οικονομικά. Τους πρόσφυγες, αυτά που συμβαίνουν εκτός συνόρων μας, στην Ουκρανία, στη Συρία. Πολλά θέματα προσυζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και ξαφνικά ένα κράτος μέλος καταφθάνει με κάποιες απαιτήσει, μεταξύ των οποίων ας επανεξετάσουμε το προήμιο της συνθήκης που αναφέρεται σε όλο και στενότερη ένωση. Αυτό οδήγησε σε κάποιο κνευρισμό, διαρωτώ με. Ήδη απαντήσατε κατά κάποιο τρόπο. Είπατε όχι, όλοι το βλέπουν αυτό με επικοδομητικό όμα. Άρα, αν κάνουμε ιστορικές συγκρίσεις, διότι είπατε ότι αυτή είναι μια περίσταση άνευ προηγουμένου, μου θυμίζει κάτι. Την κρίση της κενής θέσεως με το στρατηγό Ντεγκόλ το 1965 όπου η Γαλλία δεν ήθελε να εφαρμόσει τη διάταξη της συνθήκης για την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και μποϊκοτάρισε την Ένωση. Ε, μην πηγαίνοντα στο Συμβούλιο για ένα εξάμεινο, δεν ερχόταν καν Γάλλος εκπρόσωπος στις ε, συνεδριάσεις. Και τα άλλα κράτη-μέλη είχαν επιλογή. Θα πούμε στη Γαλλία συμμορφωθείτε, θα εφαρμοστεί η συνθήκη ω έχει και δεν κινούμεθα, δεν μετακινούμεθα, που αυτό θα προκαλούσε κρίση τέτοιου μεγέθους που θα αποχωρούσε η Γαλλία από την Ένωση τότε ή θα συνομιλήσουμε τη Γαλλία και θα συμβιβαστούμε. Κάτι που έγινε με τον περίφημο συμβιβασμό του Λουξεμβούργου που επέτρεψε να συνεχίσει η Ένωση και ο συμβιβασμός του Λουξεμβούργου τελικά λησμονήθηκε και έγινε πλέον ιστορία. Λοιπόν, υποχωρούμε για να πάρουμε φόρα για να πηδήξουμε πιο μακριά, ούτως υπήν για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το σύνολο, για να συνεχίσει να υπάρχει το σύνολο. Ίσως αυτή είναι η καλύτερη λύση. Αυτή είναι η άποψη των αλλοκατών μελών. Ποια είναι η άποψή σας από αυτό. I mean, I can't speak for the... Δεν μπορώ τώρα εγώ να πω τι σκέφτονται τα άλλα κράτη-μέλη αλλά υπάρχει νομίζω μια σεβαστή παράδοση στην Ένωση σύμφωνα με την οποία ένα κράτος μέλος ε, που έχει σημαντικά προβλήματα εισακούεται ανεξαρτήτως μεγέθους. Και έχετε δίκιο βεβαίως ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ε, είναι ο κόσμος διατεθειμένος να κάνει σοβαρές συζητήσεις για ένα προφανώς ε, σημαντικό ζήτημα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η παράδοση αυτή λοιπόν του να ακούμε και να βοηθάμε ένα κράτος μέλος ε, υπάρχει ακόμα. Και νομίζω πως είναι σημαντικό αυτό στις συζητήσεις και Ίσως γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν σοβαρές προοπτικές για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία προσεχώς θα δούμε πάντως είναι σοβαρές οι συζητήσεις με τους Βρετανούς προφανώς αλλά και με τα άλλα κράτη-μέλη Ευχαριστώ. Θα κάνω και εγώ μία ερώτηση. Κοιτάξτε, δεν στοιχηματίζω, αλλά νομίζω πως δεν έχουμε πια άλλες επιλογές. Πρέπει να συμφωνήσουμε τον Φεβρουάριο και επίσης υποθέτω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα πακέτο Το οποίο θα είναι αμοιβαία επωφελές και για όλους, ε, όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο τα κρατημέλη, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο Κομισιόν. Και αντιλαμβανόμαστε πως είναι αδύνατη η ιστορική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, οπότε η λύση θα είναι στο παράγωγο δικαίου της Ένωσης. Αυτό έχω αντιληφθεί εγώ θεωρείτε πως υπάρχει η δυνατότητα να μην υπάρχει περιθώριο κατάχρησης ε, του Βρετανικού συστήματος ε, πρόνοιας για να αντικατασταθεί η περίοδος τεσσάρων ετών που προφανώς είναι διακριτική μεταχείριση. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι οι εξής οι εγγυήσεις που είναι τόσο σημαντικές για τον κύριο Κάμερον ότι οποιαδήποτε αλλαγή της συνθήκης που ε, ε, θα πρέπει να έρθει. Μιλήσατε και για την λύση της Δανίας και για τις εγγυήσεις που παρέχει το διεθνές δίκαιο. Μπορούμε να κάνουμε κάτι ανάλογο και στην περίπτωση της Βρετανίας. Για το πρώτο που είπατε. Δεν ε, θα σχολιάσω εγώ τις ε, δυνατότητες ε, μεταρρύθμισης του Βρετανικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά γεγονός είναι πως το σύστημα κοινωνικών παραχών της Βρετανίας δεν έχει εισφορές και Τώρα πλέον θα υπάρχει το ένα ενιαίο επίδομα για όλους, ε, το οποίο παρέχεται σε εργαζόμενους όχι ανάλογα με τις εισφορές τους ε, στο σύστημα, αλλά είναι ένα αυτοδικαίωση. Και δεν νομίζω πως θα τίθεται ζήτημα να ανατραπεί αυτό. Ούτε χρειάζεται κιόλα. Ε, το σύστημα ε, είναι ως έχει, ούτως ή άλλως ε, θα το μεταρρυθμίσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά το ζήτημα το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργό ήταν το εάν ο ο αντίκτυπος ε, αυτού του συστήματος ήταν να δημιουργηθούν κίνητρα για την ελεύθερη μετακίνηση που ίσως είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά την κατάχρηση τώρα του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, κανείς δεν το θέλει αυτό. Το νομικό σύστημα της Ένωσης ε, και όλων των κρατών μελών περιέχουν ε, πολλά μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μην υπάρχει κατάχρηση του συστήματος. Θέλουμε να χρησιμοποιείται σωστά το σύστημα. Βεβαίως είναι δύσκολο να εντοπίσουμε την κατάξη, αλλά πρέπει να γίνεται. Και γι' αυτό το συζητάμε ακριβώς. Ε, τέθησαν τέτοια ζητήματα και στην επιστολή του Πρωθυπουργού. Βεβαίω ε, το θέμα αυτό αφορά ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται νομίμως ε, και πληρώνουν φόρους και το κατά πόσον μετά βεβαίω είναι δικαιούχοι. Το ζήτημα λοιπόν τώρα των συμφωνιών ε, με το προηγούμενο της Δανίας και της Ιρλανδίας δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μεταφερθεί απευθείας στην περίπτωση αυτή αλλά έχει χρησιμοποιηθεί πράγματι στο παρελθόν η απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να αποτελέσει μια συμφωνία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και μπορεί να περιγραφεί ως νομικά ζημιστική άρα. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με πλούσια νομολογία γιατί και άλλοι εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου χάνουν από καταχρήσεις. Η κυρία Κάφμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φόλ, σωστά είπατε πως έχουμε ένα περίπλοκο θέμα πολιτικό και νομικό και ελπίζουμε πράγματι να επιληθεί προς το συμφέρον της Ένωσης και της Βρετανίας μέχρι τον Φεβρουάριο. Θέλω όμως να πω πως ανησυχώ ιδιαίτερα για το εξής. Όχι μόνο λόγω του πιθανού ντόμινο, αλλά ανεξαρτήτως του εάν θα βρεθεί μια λύση η οποία θα είναι μια ειδική ρύθμιση για το Ηνωμένο Βασίλειο ή θα ισχύσει για τα 28 κράτη-μέλη και θα είναι θετική, ε, έχουμε ένα ψήφισμα όπου όλα αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν δεν θα παίξουν κανένα ρόλο. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος ε, στο Βρετανικό δημοψήφισμα. Δηλαδή αυτά τα οποία διαπραγματευόμαστε θα παίξουν, δεν θα παίξουν ρόλο στην καμπάνια γιατί γνωρίζουμε ότι έχουν μια δική τους δυναμική τα δημοψηφίσματα και το έχουμε δει και αλλού αυτό σε δημοψηφίσματα για ευρωπαϊκά ζητήματα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να εμποδίσουμε το να κάνουμε διάφορες παραχωρήσεις στη Μεγάλη Βρετανία και μετά 27 χώρες να μην έχουμε κερδίσει τίποτα γιατί δεν θα παίξει κανένα ρόλο στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια λύση. Αλλά πραγματικά κινούμαστε σε χαρτογράφη τα ύδατα και η απόφαση είναι πάλι η τελική της Μεγάλης Βρετανίας ανεξαρτήτως του τι θα κάνουμε εμείς. Ευχαριστώ. Ε, δεν μπορώ να πιθανολογήσω το πώς θα διεξαχθεί η εκστρατεία του δημοψηφίσματος για τα επιμέρους θέματα και πολύ λιγότερο μπορώ να πιθανολογήσω την έκβαση του δημοψηφίσματος. Ε, και γίνονται από πολλούς ε, ταυτόχρονες εκστρατείες. Ε, οι Πρωθυπουργοί τα έκριναν αυτά πολύ σημαντικά θέματα και φυσικά το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτό και όλοι στην Ευρώπη προσπαθούμε να ανταποκριθούμε ε, στις ανησυχίες του Πρωθυπουργού. Τώρα, το δημοψήφισμα ε, είναι θέμα του Βρετανικού λαού. Ευχαριστώ. Έρικε Γκερέρο. Ευχαριστώ. Όταν παίρνει κανείς τόσο αργά το λόγο μετά από πολλές παρεμβάσεις, ε, έχει καλυφθεί σε πολλά θέματα. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο για το οποίο μιλούμε λιγότερο στη διαδικασία αυτή. Έχουμε την εντύπωση ότι όλοι αποδέχονται αυτή την ανάγκη ε, της βελτίωσης της ενιαίας αγοράς, της ανταγωνιστικότητας. Όλα αυτά είναι σχετικά εύκολα ε, και για τη διαπραγμάτευση και για την αποδοχή. Αλλά σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές πολιτικές ε, και τις ελευθερίες, ε, οι διαπραγματεύσεις είναι πολύ πιο δύσκολες και πολύ πιο περίπλοκες. Ελάχιστο όμως λέμε για ένα τρίτο θέμα που ακροθυγώς αναφέρθηκε σε κάποια ερώτηση, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την επιθυμία του Ηνωμένου Βασιλείου να δοθούν εγγύσει ότι δεν θα αποτελέσει τμήμα καμία βελτίωση ή δεν θα συμμετέχει σε καμία ενίσχυση του γενικότερου πολιτικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, αν όντως γίνει δεκτό κάτι τέτοιο και συμφωνηθεί με συγκεκριμένους όρους, οπότε ε, επιτρέπει και σε άλλες χώρες ε, να λάβουν τέτοια θέση, δηλαδή να αναγνωριστεί και σε άλλε τέτοιο δικαίωμα εγγύηση, να μην συμμετέχουν σε ενισχυμένο πολιτικό σχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση παγώνουμε το σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη σημερινή κατάσταση. Για να μην πω ότι παλιδρομούμε. Υπάρχει ο κίνδυνο παλιδρόμηση. Ξέρω ότι δεν θα μα δώσετε πολλέ πληροφορίε, αλλά με ενδιαφέρει αν το σημείο αυτό όντω αποτελεί τμήμα τη συζήτηση και των διαπραγματεύσεων, ή μήπω οι διαπραγματεύσει εστιάζονται μόνο στο θέμα των θεμελιωδών ελευθεριών. Όχι. Ο Πρωθυπουργό ε, έδειξε τέσσερις κατηγορίες θεμάτων, όλες είναι σημαντικές και η συμφωνία μπορεί να είναι μόνο συνολική. Και Κανένα θέμα δεν ήταν εύκολο, ούτε κανένα θέμα έχει μέχρι στιγμής επιλυθεί πλήρως. Όλα είναι ανοιχτά. Και σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες σας ερωτήσεις, το θέμα της ε, όλο και στενότερης ένωσης ε, των λαών της Ευρώπης και η σχέση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και των πολλών υπόλοιπων χωρών με διαφορετικό καθεστώς ε, και με τα δικά τους εθνικά νομίσματα. Όλα αυτά τα ζητήματα άπτονται και των δικών σας, δικών σας ερωτημάτων. Και η προθυμία, η ικανότητα των κρατών μελών να συνεχίσουν στο δρόμο της ολοκλήρωσης. Δεν αμφισβητείται, κατά τη γνώμη μου, από το Ηνωμένο Βασίλειο στις συζητήσεις που γίνονται. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου και των χωρών της Ευρωσόνης, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε δημοσίω και δεν αποκαλύπτω εδώ κανένα μυστικό, δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι χώρε τη Ευρωζώνη θα πρέπει να προχωρήσουν σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση των πολιτικών του προκειμένου να δημιουργήσουν μια γνήσια και αυθεντική οικονομική και νομισματική ένωση. Και τα επιχειρήματα του Ηνωμένου Βασιλείου για το θέμα αυτό δεν αφορούν την περαιτέρω ολοκλήρωση της Ευρωζώνης, αλλά τις συνέπειες αυτής της ε, ενισχυμένης ολοκλήρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυτοεξαίρεση από το ευρώ και από τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη και δήλωσε ότι δεν έχει καμία απολύτω πρόθεση να ενταχθεί στην ε, Ευρωζώνη. Και φυσικά και το City του Λονδίνου είναι πολύ σημαντικό χρηματοπιστωτικό ε, κλάδο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και όλα αυτά αφορούν και την ε, Τραπεζική Ένωση, δεν είναι τίποτα καινούριο. Και το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να σταματήσει τους υπόλοιπους ε, να προχωρήσουν, αλλά να δουν πώς θα οργανωθούν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μορφή που έχει σήμερα και με όλη αυτή την ποικιλομορφία που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών ε, και το πώς θα εξελιχθούν περαιτέρω στο μέλλον. Υπερός Μπερές. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Τζόναθαν Φόλ, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τότε που αναλάβατε ε, την προεδρία αυτής της διαπραγματευτικής ομάδας. Το θέμα πάντως της δέσμευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της εμπλοκής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι που δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής και κατά τη γνώμη μου έχει κέρια και θεμελιώδη σημασία. Το θέμα είναι ότι χωρί αλλαγή, χωρί αναθεώρηση των συνθήκων, πολλέ από τι συνέπειε των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο για να αποτραπεί το Brexit, το οποίο και ελπίζω ότι θα αποφευθεί, θα έχει κατά πάσα πιθανότητα αντίκτυπο και στι εξουσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα συναπόφασης ή άλλα. Και φυσικά πιστεύω στην προθυμία των ε, κυβερνήσεων να καταλήξουν ε, ε, το Φεβράριο στη συμφωνία, αλλά χωρί διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώ είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Και έχω συγκεκριμένα παραδείγματα. Το δημοσιονομικό θέμα. Έχω διαβάσει αριστερά και δεξιά ότι εξαιτία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να πετύχει στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ουσιαστικά αναβάλλεται, επίσημα αναβάλλεται και ταυτόχρονα γίνεται πλήρης διαπραγμάτευσή του στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με τις υπόλοιπες χώρες και των υποχωρήσεων που θα γίνουν στην πολιτική συνοχής, τα δικαιώματα των χωρών που συνεισφέρουν και το καθεξής. Ενώ στις διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, εύλογα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησύχησε με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Γιατί διαβάζοντας τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλά σημεία που ουσιαστικά προεξοφλούσαν κάποια θέματα και στερούσαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποιες εξουσίες. Τώρα, για το θέμα του ευρώ που δεν αναφέρθηκε ακόμη και αυτό είναι κέριο ζήτημα. Και για μένα, αλλά ευτυχώ όχι μόνο για μένα. Έχω μια ανησυχία στο σημείο αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλει να επηρεαστεί από τις μεταρρυθμίσεις που ίσως χρειαστεί η Ευρωζώνη. Και φυσικά δεν θέλουμε να βρεθούμε ε, στην κατάσταση που αντιμετωπίσαμε και προηγουμένως, ώστε για να λύσουμε το υλικό πρόβλημα κοινοτοποιήσαμε ένα όργανο, ένα μηχανισμό και μάλιστα χωρίς διαβούλευση. Αυτό πάντως, πώς θα εγγυηθούμε, πώς θα δώσουμε εγγύηση ότι αυτό που θα ε, αποφασίσουμε για το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εμποδίσει την Ευρωζώνη να προχωρήσει και να κάνει αυτά που είχε αποφασίσει προς ε, το συμφέρον της Ευρωζώνης, Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και προς το συμφέρον και του Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί ο κίνδυνος ε, των, ε, αιτήσεων, των ετοιμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου σχέση με το Ευρωζώνη μου δημιουργεί φοβερές ανησυχίες. Είναι η δεύτερη συνάντηση με τον Τζόναθαν στην ΑΦΚΟ. Έχουν γίνει και άλλες συζητήσεις σε άλλες κοινοβουλευτικές συζητήσεις. Εγώ ευχαριστώ, ανταποκρίνομαι σε οποιαδήποτε πρόσκληση επιτροπής ομάδας οποτεδήποτε. Είμαι πάντα πρόθυμος να έρχομαι και το ίδιο και τα αφεντικά μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρομοίως θα εκινούντο. Ο προπολογισμό δεν συζητήθηκε σε καμία από τις διαπραγματεύσεις που συμμετείχα. Δεν αναφέρεται στην επιστολή του Πρωθυπουργού. το θέμα της περαιτέρω πρόοδου της Ευρωζώνης. Δεν είδα πουθενά να υπάρχει ισχυρισμό σύμφωνα με τον οποίο η οδήποτε μέρος θέλει αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων να είναι παρεμπόδιση αποφάσεων της Ευρωζώνης για περαιτέρω ολοκλήρωση. δεν βλέπω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλα κάτι μέλη να το δέχονται αυτό. Δεν πιστεύω ότι αυτό ήταν πρόθεση της ε, Βρετανικής κυβερνήσεως. Αφορά τη διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ χωρών Ευρωζώρης και των άλλων στην κοινή ενή αγορά δεν είναι νέο ζήτημα στις συζητήσεις περί τραπεζικής στις οποίες συμμετείχε και το Ευρωκοινοβούλιο, αυτά τα θέματα ανελήφθησαν ενδελεχέστατα και η χρήση του προπολογισμού, όπως αναφέρατε, στην περίπτωση της Ελλάδας και λύθηκε αυτό και των ισχυρισμών ε, περί ε, διακρίσεων στον αφορά το νόμισμα ή την τοποθεσία. Αυτά τα θέματα επελήφθησαν, επελήφθησαν στην Τραπεζική Ένωση τις σχετικές συζητήσεις Δημιουργείται έτσι μια βάση επί της οποίας μπορούν να ε, ευρεωθούν αρχές και ελπίζω το θέμα να επιληθεί με έναν τρόπο ικανοποιητικό για όλα τα μέρη. Είναι ευαίσθητο θέμα, σημαντικό, αλλά δηλώνω σαφέστατα ότι έχω την εντύπωση ότι πραγματικά κανείς δεν επιδιώκει να χρησιμοποιήσει το θέμα αυτό ως τρόπο παρεμποδίσεως ιονδήποτε μελλοντικών αποφάσεων σχετικών με τη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Ο Ραμόν Χαουρέκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δύο ρωτήσεις ε, συντομότατες όσον αφορά τον χρονισμό και την όλη διαδικασία. Όσον αφορά τον χρονισμό, το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να κάνει το δημοψήφισμα ε, εάν υπάρξει συμφωνία του επόμενου μήνες. Θα γίνει το δημοψήφισμα πιστεύετε φέτος. Αν όχι, μέχρι πότε ε, θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Θεωρείτε ότι μπορούν να παραταθούν οι διαπραγματεύσεις φέτος. Δεύτερη ερώτηση. Από τη στιγμή που θα υπάρξει μια συμφωνία στο Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προβεί σε μεταρρυθμίσεις. Ενδεχομένως, διότι ο Κάμερον θα ήθελε μια συμφωνία αμετάκλητη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο οι μεταρρυθμίσεις μας να είναι συνέπεια του Βρετανικού ναι. Δηλαδή, αν εμείς κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που μας ζητάει η Μεγάλη Βρετανία και μετά στο δημοψήφισμα υπάρξει αποτέλεσμα αρνητικό, θα, δεν θα είναι λογικές οι μεταρρυθμίσεις θα υπάρξει πολιτική συμφωνία ε, να γίνουν μεταρρυθμίσεις ε, αμετάκλητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει νέο Βρετανικό. Δηλαδή το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συζητήσει μεταρρυθμίσεις επί τη βάση της αποφάσεως που θα ληφθεί στην ε, Βρετανία. Να παραμείνει στην Ένωση. Έτσι έχουν τα πράγματα. Απάντηση. Ο χρονισμός αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Η μόνη βεβαιότητα είναι ότι το δημοψήφισμα θα λάβει χώρα πριν το τέλος του 2017. Μπορεί να λάβει χώρα πριν. Και θα πρέπει να δούμε όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, όποτε γίνει αυτό, τότε ο Πρωθυπουργό και η Βρετανική κυβέρνηση θα αποφασίσουν τα δέοντα. Εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τη διαδικασία. Δεν μπορώ να σχολιάσω, ούτε θέλω να προβώ σε εικασίες για τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Θα είναι μια δημοκρατική διαδικασία μετά από εκστρατεία, προεκλογική, ψηφοφορία θα λάβει χώρα και αυτό αφορά το βρετανικό λαό. Και εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω ο ίδιος γιατί έχω ζήσει στο εξωτερικό επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν θέλω τώρα να προβώ σε εικασίες για δεχόμενες συνέπειες ε, της αποφάσεως είτε ναι είτε όχι στις διαδικασίες που ήδη θα έχουν ε, δρομολογηθεί. Συγγνώμη, ο Πάλο Ράντζο, πολύ σύντομη ερώτηση, αν επιτρέπετε. Και ο Ραμόν θέλει να συνεχίσει. Θα συνεχίσει. Δεύτερη ερώτηση, λέει ο Ραμόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέτασε τη δυνατότητα οι μεταρρυθμίσεις ε, που χρειάζονται στην ένωμη μας τάξη να γίνουν μετά το δημοψήφισμα, όχι πριν. Το εξέτασε καθόλου αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Κοιτάξτε, δεν ε, εξετάζουμε ποια θα είναι η επιρροή του αποτελέσματος θα δούμε τι θα γίνει όποτε διεξαχθεί το δημοψήφισμα. Τότε θα δούμε πώς θα επηρεάσει τα πράγματα το αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να κρατήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι είναι υποφελές για την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι τέτοιο. Και χωρίς η αδίποτε παρέμβαση πιστεύουμε ότι είναι και προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά είχα με ένα κατεπήγον πρόβλημα στην Προεδρία του ΕΡΚ να επιλύσω. Συντομότατο ερώτημα. Θα ήθελα να ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν διαπραγματεύεται, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δηλαδή, λαμβάνει υπόψη το εξή. Κάποιες παραχωρήσεις που το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στη, όσον αφορά τη θέση άλλων κρατών μελών στο μέλλον. Να δημιουργηθεί κάποια ασύμετρη σχέση. Όταν διαπραγματευόμεθα εν ονόμα της Ευρωπαϊκής με το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε επίγνωση ότι αυτό μπορεί να έχει κάποιες συνέπειες για άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν είναι το ερώτημα. Απάντηση ναι, ναι, Βεβαίω. Και τα άλλα κράτη-μέλη υπήρξαν σαφέστατα μας εξήγησαν, όπως τα εξήγησαν και στους Βρετανούς, είμαι σίγουρος, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αυτών των θεμάτων, ποιος θα ήταν, ποιος είναι για αυτές τις χώρες. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε αυτή τη συζήτηση. Θέλω να πω ότι ελπίζω τελευταία συζήτηση, την επόμενη φορά που θα έρθετε θα παρουσιάσετε τα αποτελέσματα. Ας ελπίσουμε ότι Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου ή και μετά το Πάσχα, το δεχόμαστε και αυτό, θα μας δώσετε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στις διαπραγματεύσεις. Thank Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ. Θα ήθελα να συνεχίσουμε. Ε, Ρίκη Γιολάινε, παρακαλώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, Υπουργό Μπέρτ Κούντερς, που είναι ο Ολλανδός ε, Υπουργός ασκών την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντική η Ολλανδική Προεδρία και για τη δική μας ε, Επιτροπή. Περιμένουμε πολλές χαρμόσυνες ε, ειδήσει από εσά. Ξέρω ότι έχετε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα σήμερα και κάποιες ε, επιτροπές πολύ πιο δύσκολες από τη, δικές, από τη δική μας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω εγκάρδια, να σας ευχηθώ καλή τύχη, καλή επιτυχία στην Ολλανδική Προεδρία και να σας δώσω και το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που επιστρέφω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είστε το μοναδικό έρετο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο και εδώ πέρα λαμβάνουν χώρα σημαντικές ε, συζητήσεις και υπάρχει και ουσία εκτός από την πολιτική και βέβαια υπάρχει και η συζήτηση για τα θεσμικά ζητήματα της Επιτροπής σας που είναι πάρα πολύ σημαντική. Η τελευταία μας Προεδρία ήταν το 2004 και πολλά άλλαξαν έκτοτε και για το Κοινοβούλιο και έχω δει πως ε, εξελίχθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πραγματικό συνομοθέτη που είναι σήμερα. Σκοπεύουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας να εντείνουμε τις καλές σχέσεις που έχουμε και την συστηματική στρατηγική μας ε, συνεργασία και αναμένουμε μια στενή ε, συνεργασία όπως σας είπα. Γι' αυτό ακριβώς ε, θα εκπροσωπήσω το Συμβούλιο μαζί με την Ζανίν ε, την Υπουργό Άμυνας που θα την θυμάστε αρκετοί από εσάς, ήταν Ευρωβουλευτής Τώρα, πριν αναφέρω τις προτεραιότητες της Προεδρίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία του Λουξεμβούργου. Νομίζω πως θα μιλήσετε και με τον Υπουργό Σμιτ ε, το απόγευμα. Να τους συγχαρώ λοιπόν για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν ε, και τον κύριο Υπουργό. Αναλαμβάνουμε και είναι σαφές νομίζω την Προεδρία του Συμβουλίου σε δύσκολες συνθήκες συνθήκες που καθιστούν ξεκάθαρη την αναγκαιότητα της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξτρεμισμό, μετανάστευση, οικονομική ανασφάλεια πολλών πολιτών και μια δύσκολη κατάσταση στα ανατολικά μας σύνορα. Οπότε η Προεδρία αυτή δεν θα αντιμετωπίσει μόνο τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει εμείς στην στρατηγική μας ατζέντα, αλλά θα υπάρχουν πολλοί άγνωστοι παράγοντες, πράγματα που ξέρουμε ότι είναι άγνωστα και πράγματα που δεν ξέρουμε ακόμα. Και βεβαίως υπάρχει και ζήτημα εμπιστοσύνη μεταξύ χωρών και εντός των χωρών. Και αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος ε, περιμένει λύσεις από την Ευρώπη και δικαίως γιατί τα τρία ζητήματα που ανέφερα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνο σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως έχει έτοιμες απαντήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Γι' αυτό ακριβώς ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, πέρα από οράματα και ιδέες, χρειαζόμαστε και εσάς ως εταίρους, έτσι ώστε η Ευρώπη να ανταποκριθεί στην υπόσχεσή της για ένα καλύτερο μέλλον για όλους ε, τους Ευρωπαίους. Είμαι σίγουρος πως οι Ευρωπαίοι έχουμε το μυαλό και την θέληση και τους ανθρώπους για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Ε, το κάναμε και στο παρελθόν. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι σκληρή δουλειά, ψυχραιμία, επιμονή και μεγάλη καρδιά. Θεωρούμε πως είναι δυνατόν αυτό. Εμείς θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς ε, διαμεσολαβητές, αλλά βεβαίως μιλάμε για το μέλλον της χώρας μας και των χωρών σας. Δεν είμαστε ουδέτεροι. Θέλουμε να επιτύχουμε και θα είμαστε και ρεαλιστές αυτό το οποίο χρειάζεται τώρα η Ευρώπη είναι απτά αποτελέσματα για τα πράγματα που μόλις ανέφερα. Στο πλαίσιο λοιπόν της ε, στρατηγικής ατζέντα ε, και των γνωστών και αγνώστων πραγμάτων που είπα, θα εστιάσουμε στις ε, προτεραιότητες πολιτικής μας. Η Ευρώπη που θα δημιουργεί δουλειές και θα καινοτομεί μια συνολική αντιμετώπιση της ε, μετανάστευσης και της ε, διεθνούς ασφάλειας ε, που συζήτησα σε μια άλλη επιτροπή και βεβαίως υγιή δημόσια οικονομικά και μια πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια. Θα ήθελα λοιπόν να παρουσιάσω κάποια ζητήματα σημαντικά για τη δική σας επιτροπή. Με βάση τις προκλήσεις που ανέφερα, πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε τις ε, διασυνδέσεις μεταξύ των ε, θεσμικών κρατών των ε, μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών λαών καθώς διακυβεύεται αυτή τη στιγμή η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων. Πάρα πολλοί άνθρωποι και νοικοκυριά και παρτεύουσες ασκούν κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά εξίσου πολλοί αντιλαμβάνονται πως κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μόνος του και υπάρχουν περισσότερα στοιχεία που μας ενώνουν από όσα μας χωρίζουν. Η δυσαρέσκεια όσον αφορά την ανικανότητα των 28 κρατών μελών οδηγεί σε ευρωσκεπτικισμό, οπότε θα πρέπει να βρούμε τον βέλτιστο συνδυασμό ελευθερίας των κρατών μελών να χαράξουν την πολιτική τους, αλλά και παροχής λύσεων. Και πρέπει να διασφαλίσουμε πως θα είμαστε αποφασιστικοί, αλλά να αναγνωρίσουμε και την προσέγγιση των πολιτών μας. Θεωρούμε λοιπόν πως εδώ έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, να ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και τον διάλογο μεταξύ Κοινοβουλίων και Κοινοβουλίου και Κομισιών. Όταν μιλάω με Εθνικά Κοινοβούλια, καμιά φορά μου λένε ε, ότι δεν ενδιαφέρεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόλου. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό ισχύει και ούτε θεωρώ πως υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός. Ναι, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ειδικά στα συνταγματικά ζητήματα, αλλά εκπροσωπείτε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους και μπορείτε να διαμορφώσετε τον Δήμο που χρειάζεται να έχουμε πολίτες και όχι μόνο καταναλωτές ε, και να έχουμε μια κοινή κυριαρχία και άρα μια δημοκρατία. Στα διεθνή τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια από τα ζητήματα που θα σας απασχολήσουν νομίζω. Πρώτα απ' όλα για την ε, διοργανική συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Νομίζω πως αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όλοι γνωρίζουμε πως είναι πιο ε, σημαντικό από όσο είναι ενδιαφέρον. Και πάρα πολλοί στο Κομισιόν και στο Συμβούλιο είπαν πως ποτέ δεν θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο και όμως εδώ είμαστε οι κύριοι Φερχόφστατ, Σμιτ ε, και Τίμερμανς ε, και αξίζουν τον σεβασμό μας και πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για καλύτερη νομοθεσία και περισσότερη διαφάνεια και ίσως βεβαίως ε, οι νομικές λεπτομέρειες να φαίνονται περίεργες αλλά πρέπει να προχωρήσουμε για να λειτουργήσει η υπόθεση και αν ακούγεται ως κάτι το τεχνικό, η διοργανική συμφωνία έχει μεγάλη σημασία για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχύσουμε την ε, νομοποίηση της Ένωσης και να επιτύχουμε αποτελέσματα και ζητάω και από εσά και από μας να την κυρώσουμε το συντομότερο δυνατόν και να αρχίσει να λειτουργεί. Θέλουμε να εστιάσουμε στην εφαρμογή της ε, κατά την διάρκεια της ε, Προεδρίας μας, να συνεχίσουμε τη δουλειά που έκανε το Λουξεμβούργο, να εφαρμοστούν οι αρχές της ε, στο δεύτερο μισό της θητείας της Επιτροπής. Αυτό είναι σημαντικό και για τα τρία θεσμικά όργανα. Η εφαρμογή της Διοργανικής Συμφωνίας σημαίνει πως το Συμβούλιο θα πρέπει να σκεφτεί τις εσωτερικές του διαδικασίες, ειδικά όσον αφορά την προετοιμασία του ετήσιου προγράμματος εργασίας της ε, Κομισιόν. Χρειαζόμαστε μια διαδικασία αξιόπιστη και σε αντίθεση με το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα ορίσει διαδικασία. Πρέπει να συνεργαστούμε και στην κοινή εφαρμογή του προγράμματος της Κομισιόν όταν υιοθετηθεί. Επίσης, το Συμβούλιο θα πρέπει να σκεφτεί το πώς χρησιμοποιεί τα μέσα για την καλύτερη νομοθεσία, αξιολόγηση αντικτύπου, διαβουλεύσεις ε, και αξιολογήσεις, δύσκολες λέξεις, ε, εκτός αυτές τις αιθούσης ίσως ακατανόητες, αλλά πάρα πολύ σημαντικές. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα εντός του Συμβουλίου και σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και η Προεδρία μας ε, το θεωρεί ως κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Θα συνεργαστούμε με εσά και την Κομισιόν ε, για τις ε, διατάξεις, ε, για τη διαφάνεια, για το συντονισμό της νομοθετικής διαδικασίας και πρέπει νομίζω να αναβιάσουμε την κοινή διοργανική ομάδα και αναμένουμε να ολοκληρωθούν σύντομα οι διαπραγματεύσεις αυτές τους επόμενους μήνες. Για την διαφάνεια τώρα θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε αυτό το κομμάτι της ε, διοργανικής συμφωνίας. Όλοι συνειδητοποιούν πως υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της ε, δημοκρατικής νομοποίησης και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης και εδώ πέρα πραγματικά πρέπει όλοι μας να είμαστε ανοιχτοί. Κατά τη διάρκεια της ε, προεδρίας μας ε, θα προωθήσουμε την περισσότερη διαφάνεια στην λήψη αποφάσεων. Υπάρχουν τρόποι να γίνει αυτό σε διάφορες τομείς. Η συμφωνία TTIP είναι ένα καλό παράδειγμα όπου έχει μεγάλη σημασία η διαφάνεια. Αν θέλουμε τη στήριξη της κοινή γνώμης πρέπει να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση για το θέμα αυτό Ευτυχώς πολλά πράγματα έχουν γίνει ήδη όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για την TTIP. Ένα άλλο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ο κώδικας συμπεριφοράς. Το Συμβούλιο εξετάζει σοβαρά το ζήτημα της ε, διαφάνειας ε, των εγγράφων του Συμβουλίου πέρα από συγκεκριμένους ε, τομείς απαιτείται και μια συστηματική αντιμετώπιση της διαφάνειας χρειάζονται καφείς διαρθρωτικές αλλαγές όχι επανάσταση να δούμε, κάνουμε απλά κάποια συγκεκριμένα εστιασμένα αναγκαία βήματα και αυτά θέλω να τα κάνουμε μαζί σας. Άρα είμαστε ικανοποιημένοι στις συμφωνίες που έγιναν στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Δείχνει πως και τα τρία θεσμικά όργανα θέλουμε να βελτιώσουμε τη διαφάνεια της Ευρώπης και οι συμφωνίες αυτές θα είναι το πρώτο σημείο αφετηρίας. Π.χ η συμφωνία για τη διαφάνεια των διαλόγων, των τριμερών διαλόγων. Ένα ευαίσθητο ζήτημα, όπου βεβαίω πρέπει να βρούμε την ισορροπία με την αποτελεσματικότητα που πρέπει να έχουμε. Πρέπει να το δούμε πάρα πολύ προσεκτικά, οπωσδήποτε στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασία, να αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου σε τακτική βάση για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τον ρόλο μας ως συνομοθέτες. Πέρα από αυτό πρέπει να συνεργαστούμε για μια κοινή βάση δεδομένων που θα είναι χρήσιμη για τους ε, χρήστες που δεν είναι ειδικευμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως ε, να ανταποκριθούμε σε αυτά τα οποία αναφέρουν οι διατάξεις για την ίχνη λασιμότητα και ο πρόεδρος Γιούνκερ μίλησε για ένα υποχρεωτικό μήτρο στις πολιτικές του προτεραιότητες και το πρόγραμμα εργασίας κομισιών για το 2016 και αναμένουμε τις προτάσεις με μεγάλο ενδιαφέρον. Εάν η Κομισιόν βεβαίως φέρει μια πρόταση για ένα υποχρεωτικό μητρό το επόμενο εξάμεινο, οπωσδήποτε η Προεδρία μας θα αρχίσει αμέσως τις διαπραγματεύσεις. Θα αναφερθώ τώρα στη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Εκλογικού Νόμου τα τελευταία χρόνια βλέπουμε χαμηλή προσέλευση στις ε, εκλογές ε, που είναι ο άμεσος τρόπος για να εκφράσουν οι πολίτες την άποψή τους και κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον των πολιτών. Το Συμβούλιο συμφωνεί με αυτή την ε, φιλοδοξία του Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου. Επίσης είχαμε μια μεγάλη συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Έχουν γίνει κάποιες ανταλλαγές απόψεων που κατέστησαν σαφές πως και εντό του Συμβουλίου ίσω υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτόν τον κοινό στόχο. Αυτό δεν ισχύει νομίζω λιγότερο εντός του Κοινοβουλίου από ότι εντός του Συμβουλίου. Σημειώσαμε τα όσα είπατε στην πρότασή σας και η Προεδρία μας θα ξεκινήσει επίσημες συζητήσεις στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου με βάση τη δική σας πρόταση του Κοινοβουλίου. Όμως ε, βεβαίως υπάρχουν διαδικαστικές υπάρχουν διαδικαστικά, διαδικαστικοί περιορισμοί στο εθνικό επίπεδο καθώς πρέπει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει όλων των κρατών μελών και βεβαίως ε, θα ενημερώσουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο των συζητήσεων μόλις ε, έχουμε κάποια αποτελέσματα των συζητήσεων. Κάτι άλλο βεβαίως ε, το οποίο αφορά το δικαίωμα της εξέτασης πρέπει να λειτουργούν δημοκρατικά τα θεσμικά όργανα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι των εποπτικών αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο και όπως ξέρετε το Συμβούλιο έχει κάποιες ε, θεμελιώδεις νομικές και θεσμικές επιφυλάξεις. Ομόφωνα το Συμβούλιο θεωρεί πως είναι τόσο σοβαρά τα ζητήματα ώστε θα πρέπει να είναι εκτός των διαπραγματεύσεων Είμαστε βεβαίως και καλωσορίζουμε ε, την ε, πρόθεση του εισηγητού να δεχτεί κάποιες από τις ανησυχίες του Συμβουλίου και επαναλαμβάνουμε την θέλησή μας να συνεργαστούμε επικοδομητικά με το Κοινοβούλιο και βεβαίως αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσετε τις ε, ανησυχίες μας. Και σκοπεύουμε να συναντηθούμε και με τον εισηγητή για να δούμε τι θα ε, κάνουμε με τον φάκελο αυτόν. Η πρωτοβουλία των πολιτών. Όπως ανέφερα πριν, ε, η σύνδεση με τους πολίτες είναι απολύτως απαραίτητη για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι ένα σημαντικό μέσο έτσι ώστε οι πολίτες να μιλήσουν άμεσα και να έρθουν πιο κοντά στην Ένωση, όμως ο χαμηλός αριθμός επιτυχημένων πρωτοβουλειών δείχνουν πως τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή έχουν κάποιες ελλείψεις και χρειάζονται βελτίωση για να λειτουργήσουν καλύτερα. Καλώς ορίζουμε τα βήματα που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση από την Κομισιόν για να αξιολογήσουμε την εφαρμογή του σχετικού κανονισμού και καλωσορίζουμε τη δουλειά που έχει κάνει ο κ. Σέφλιν εδώ πέρα και αναμένουμε τις ε, περαιτέρω διαβουλεύσεις της Κομισιόν για να βελτιωθεί αυτό το σύστημα για να εγγυηθούμε ότι θα έχουμε ένα αποτελεσματικό μέσο για την Ευρωπαϊκή Συμμετοχική Δημοκρατία. Για να καταλήξω, για να ακούσουμε μετά και τις δικές σας απόψεις. η Προεδρία αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη υπόθεση. Πάντα βεβαίω είναι, αλλά τώρα έχουμε κάποιες προκλήσεις όσον αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως το ότι έχουμε επιτύχει. Είμαστε η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον πλανήτη. Έχουμε μια ειρήνη. Μια ήπειρο ειρηνική. Τα παιδιά μας πάνε σχολείο. Έχουμε καθαρό αέρα. Φροντίζουμε τους ηλικιωμένου εντό ε, των συνόρων μα γίνεται σεβαστή η δημοκρατία και οι μειονότητε, αν και βλέπουμε πολλές συζητήσεις ω προ αυτό και ε, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε και στο παρελθόν βλέπουμε πω ε, όσοι δεν τα έχουν αυτά διακινδυνεύουν τι ζωέ του για να τα αποκτήσουν. Γι' το ευρωπαϊκό όνειρο είναι κάτι το πραγματικό και ελπίζω πω θα τα εγγόνια μας ε, θα μιλάνε σε 50 χρόνια για την περίοδο αυτή όταν η Ευρώπη ανταποκρίθηκε στις ε, δυσκολίες ε, ότι δεν ήταν μόνο μία οργάνωση και ένας οργανισμός καλού καιρού αλλά ένας οργανισμός παντός καιρού και θεωρώ πως τα καλύτερα έρχονται θα ε, εργαστούμε λοιπόν σκληρά, να είμαστε ένας αξιόπιστος εταίρος ε, για να μπορέσουμε να λάβουμε σκληρές αποφάσεις και να εφαρμόσουμε σοβαρές μεταρρυθμίσεις όπου αυτό απαιτείται. Καμιά φορά αυτό σημαίνει περισσότερη Ευρώπη, καμιά φορά λιγότερη, αλλά πάνω απ' όλα ελπίζω καλύτερη Ευρώπη. Μια ένωση που θα έχει αποτελέσματα, θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις μελλοντικέ προκλήσεις και θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών της. Νομίζω πως η Ευρώπη πρέπει να ξαναβρει λίγο έτσι, το ρυθμό της και αναμένω τη συνεργασία μαζί σας κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την ε, γνωστή παραδοσιακή για την Ολλανδία ε, προθυμία, ειλικρίνεια. Ε, ήσταν πραγματικά πολύ ντόμπρος. Μας παρουσιάσατε όλα αυτά τα θέματα και βάλατε και τα συνταγματικά ζητήματα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το πλαίσιο των προτεραιοτήτων και των στόχων τη Ολλανδική Προεδρία. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και χρήσιμο για τη συζήτηση και ευελπιστούμε ότι ε, θα βοηθήσει αυτή η προσήλωση που δείχνεται και στα θέματα που μας είναι προσφυλή, ώστε να έχουμε αποτελέσματα για αυτά στη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους, πρώτα στο Ιω Λάινεν και μετά στο Τζορτ Σέμπλινγκ. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, σας ευχαριστώ για αυτό το οποίο μας είπατε. Τα πολύ ικανοποιητικά για μια ισχυρή Ευρώπη που θα είναι δημοκρατική και κοντά στους πολίτες. Τελευταία Ολλανδική Προεδρία ήταν το 2004, ωραίες εποχές το κλίμα ήταν θετικό, είχαμε μπροστά μας τη διεύρυνση, όλοι ήταν ενωμένοι, σήμερα είναι αλλιώς τα πράγματα. Το είπατε και η επόμενη προεδρία θα είναι το 2028-29. Και πράγματι θα δούμε τι θα λένε τότε οι άνθρωποι για εμάς, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ο κίνδυνος να διαλυθούμε και θεωρώ πως ε, το εξάμεινο το δικό σας ε, θα αποτελέσει ένα τεστ συνοχής για την Ευρωπαϊκή Ένωση αν θα ξαναπάμε σε ε, εθνικισμούς που θα μας διχάσουν και αυτός ο κίνδυνος ισχύει για τα πάντα όχι μόνο για το Βρετανικό δημοψήφισμα αλλά και για το τι συμβαίνει στην Πολωνία και σε άλλες χώρες όπου δεν έχουμε πια τις ίδιες αξίες αλλά κυλάμε σε εγωιστικά εθνικά συμφέροντα. Αναφέρατε κάποια ζητήματα, κάτι δεν άκουσα όμως. Η πρόταση του Κοινοβουλίου για να βελτιωθούν οι επόμενες ευρωεκλογές. Μιλήσατε για δημοκρατία, για Ευρώπη των πολιτών. Οι ευρωεκλογές είναι κάτι το μοναδικό και γνωρίζουμε πως ε, έχουμε πολλά ελλείμματα ακόμα και πρέπει να ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα για να γίνουν πιο ελκυστικές για να υπάρχει μια ευρωπαϊκή διάσταση εκτιμώ λοιπόν πάρα πολύ για τη μεταρρύθμιση των ευρωεκλογών χρειαζόμαστε λοιπόν ένα, ένα αποτέλεσμα στο τέλος αυτού του έτους γιατί σε κάποιες χώρες θα πρέπει να αλλάξουν οι νομοθεσίες και αν γίνει αυτό να προλάβουν το 2019 πρέπει να βιαστείτε. Εγώ είμαι εισηγητής για την ομάδα μου και για την πρωτοβουλία της διαφάνειας. Εδώ και χρόνια αναρωτιόμαστε γιατί δεν μπορεί να συνεισφέρει στο Μητρό Διαφάνεια στο Συμβούλιο. Νομίζω είναι ένα θέμα αυτό το έφυξε η η Προεδρία στην ομάδα εργασίας, δηλαδή να έχουμε ένα κοινό μητρό διαφάνειας και των τριών θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, θέλετε να απαντάτε ξεχωριστά σε κάθε ομιλητή ή θέλετε να συγκεντρώσουμε μερικές ερωτήσεις πρώτα. Να συγκεντρώσουμε. Ωραία. Ο Τζόρτζ Σέπφλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να σας καλωσορίσω κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και εκ μέρους του ΕΛΚ στην Επιτροπή μας. Ήταν ε, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η επισκόπηση που μας κάνατε. Καλύψατε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ε, και μάλιστα θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις ε, σε στρατηγικό επίπεδο. Κάτι βραχιοπρόθεσμο που δεν αναφέρατε, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι τι συμβαίνει σε σχέση ε, με τις διαπραγματεύσεις ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο και την επικείμενη διάσκεψη κορυφής. Έχετε κάτι ιδιαίτερο να μας πείτε, κάτι καινούριο μπορείτε να προσθέσετε ενδεχομένω σε αυτά που μας είπατε. Άλλο θέμα, μετανάστευση. Ποιες είναι οι στρατηγικές σας σκέψεις ε, σε θέματα κανονισμού του Δουβλίνου. Ξέρετε ότι είμαι Ούγγρος, οπότε είμαστε σχεδόν στα εξωτερικά σύνορα και γνωρίζετε ότι περιμένουμε ως ονούπο νέα μεγάλη ροή προσφύγων και μετακινούνται όλο και περισσότερο προς τα βορρά. Στρατηγικά πώς θα τα βλέπετε όλα αυτά, τι μέτρα μπορούν να θεσπιστούν. Από αυτά που έχω διαπιστώσει εγώ τουλάχιστον, τα μέχρι τώρα μέτρα δεν έχουν λειτουργήσει και πολύ αποτελεσματικά την απάντηση την αφήνω σε εσά πάντω. Ένα άλλο συναφέ θέμα με το προηγούμενο είναι το εκόλουθο. Υπάρχει, υπάρχουν κάποιες προτάσεις για την ε, διαφύλαξη της ασφάλειας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή η παροχή ασφάλειας είναι από τις ε, πρωταρχικές λειτουργίες και υποχρεώσεις του κάθε κράτους. Βέβαια, το ε, πρόβλημα πια είναι πανευρωπαϊκό. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει ένα είδο ε, ανταλλαγή πληροφοριών ε, για να δοθεί και μια πιο ευρωπαϊκή λύση σε αυτή την εξασφάλιση τη ασφάλεια. Χαιρόμαστε για αυτά που είπατε για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών και συμφωνώ μαζί σα ότι δεν ήταν λαμπρή επιτυχία μέχρι στιγμή αυτού του μέτρου και φαντάζομαι το γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε οι βελτιώσει που αναφέρατε πού ακριβώς θα κατευθυνθούν. Και κάτι άλλο που θα γνωρίζετε κι εσείς είναι ότι έχουμε σημαντική και αυξανόμενη δυσαρέσκεια των μη κυβερνητικών οργανώσεων και το, της κοινωνίας των πολιτών για το θέμα αυτό. Δεν λέω ότι είναι το πιο καταπήγον ζήτημα, αλλά αν λάβουμε υπόψη το θέμα της επαφής ανάγκης δημιουργίας δεσμών και της εμπιστοσύνης ανάκτησης εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών και το θέμα του Ευρωπαϊκού Δήμου. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών είναι πολύ σημαντικό μηχανισμό και σε αυτό το πλαίσιο. Και τέλο, μιλήσατε για τι σχέσει με τα εθνικά κοινοβούλια. Πιο συγκεκριμένα, πώ βλέπετε τι σχέσει με τα εθνικά κοινοβούλια. Ξέρω ότι είναι δύσκολο το θέμα, γιατί υπάρχουν συμφέροντα από όλων των πλευρών και δεν είναι εύκολο να το συμφιλιώσουμε πολλές φορές. Έχετε να προσθέσετε τίποτα για τη σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ακούσουμε και τον Ραμό Χαουρέγγι και μετά θα δώσω τον, πρόεδρο, τον λόγο στον Υπουργό για να απαντήσει. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Εγώ είμαι ο εισηγητής για το δικαίωμα εξέτασης ε, που αναφέρατε κι εσείς στην ε, εισαγωγική σας ομιλία. Σας ευχαριστώ θερμά για τα λόγια σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να θέσετε ως στόχο της Προεδρίας, της Ολλανδικής Προεδρίας, την επίλυση αυτού του προβλήματος, που πραγματεύεται και η δική μου έκθεση για το δικαίωμα εξέτασης, right of inquiry. Και μάλιστα είχατε συνάντηση με την πρόεδρο μας, την Τανούτα Χιούμπνερ, και εκρεμεί και το θέμα της ε, μεταγενέστερης ε, συνάντησή μα για το θέμα αυτό. Πάντω, σα ευχαριστώ για την προθυμία και την καλή βούληση που δείξατε. Και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι μιλούμε για ένα θεμελιώδε ζήτημα, για ένα θέμα κλειδί τη ίδια τη φύση ε, του Κοινοβουλίου. Και όπω είπατε, το Κοινοβούλιο μα είναι ένα πραγματικό κοινοβούλιο, ένα γνήσιο κοινοβούλιο με όλο και περισσότερε νομοθετικέ αρμοδιότητε. Και η κοινοβουλευτική λειτουργία όλων των κοινοβουλίων του κόσμου ε, περιλαμβάνει τον έλεγχο, τον έλεγχο της κυβέρνησης, ε, το, την νομοθετική λειτουργία αλλά και την εκπροσώπηση των Ευρωπαίων πολιτών. Όλα αυτά τα στοιχεία ανήκουν στον πυρήνα της κοινοβουλευτικής λειτουργίας και δεν είναι τυχαίο που η συνθήκη της Λισαβόνας εκχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας ε, και μαζί με τον εκλογικό νόμο οι μόνοι τομείς στους οποίους έχουμε δικαίωμα πρωτοβουλίας είναι αυτή και μας έδωσε και τη δυνατότητα να εκπονήσουμε ένα κανονισμό με θέμα το δικαίωμα εξέτασης και τις ε, εξεταστικές των πραγμάτων επιτροπές ή τις ερευνητικές επιτροπές. Βέβαια είναι κάπως ε, άβολη αυτή η εξουσία που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα κράτη-μέλη. Και μάλιστα πρόσφατα διαπιστώσαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκοπεύει να στήσει και μια νέα εξεταστική επιτροπή για το θέμα της Volkswagen. Και φυσικά τα κράτη-μέλη έχουν θορυβηθεί, γιατί δεν ξέρουν ποια θα είναι τα δικαιώματα εξουσίας αυτές της Εξεταστικής Επιτροπής, ποιους υπουργούς θα καλέσει και στα Ισπανικά έχουμε μία έκφραση, δεν ξέρω αν υπάρχει και στα Ολλανδικά κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά σαν καυτή πατάτα είναι σαν να βάζει κανείς το χέρι του στη φωτιά. Γι' αυτό και θα ήθελα να σας εκφράσω εδώ την δυσφορία μου, γιατί ένα χρόνο επιχειρώ ε, μία συνομιλία με το Συμβούλιο και δεν τα κατάφερα. Είχαμε και ένα έγγραφο εργασίας για να δείξουμε την ε, επιθυμία μας να αναθεωρήσουμε το προηγούμενο κείμενο και να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα εξάμεινο ε, προσπάθησα μάταια με τη Λετανική Προεδρία να κινήσω το θέμα. Το ίδιο και με τον κύριο Σμιτ πριν από ένα εξάμεινο, Λουξεμβουριανή Προεδρία. Το Σεπτέμβριο του 2015 μου υποσχέθηκε συνομιλίες και λίγο μετά στο Στρασβούργο του πρότεινα να τροποποιήσουμε το κείμενο και του εξήγησε ότι είναι απόλυτα πρόθυμο. Σίγουρα το Συμβούλιο δεν είναι πρόθυμο και δεν του αρέσει το κείμενο. Ήταν αδύνατον να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για συνάντηση με το Συμβούλιο. Πραγματικά αισθάνομαι μεγάλη απογοήτευση, εκνευρισμό, αλλά έχω και μεγάλε προσδοκίε από την Ολλανδική Προεδρία. Ελπίζω ότι θα επιλύσουμε το πρόβλημα και πραγματικά δεν θέλω να γνωρίζετε ότι είμαστε απόλυτα πρόθυμοι και εγώ και η πρόεδρός μας η Ντανίτα Χιούμπνερ θα σταθούμε στο πλευρό σας και θα σας αποδείξουμε ότι είμαστε πρόθυμοι και έχουμε τη βούληση να σημειώσουμε πρόοδο. Αλλά σας θέλουμε παρακαλώ, να ξεκινήσουμε επιτέλους τις συζητήσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις ε, που μου θέσατε. Προς τον κύριο Λάινε να πω τα καταρχάς, δεν ξέρω τι θα πούμε στο μέλλον, 2027-2009. Αυτό που είδα από το 2004 που είχαμε την Προεδρία, είδα βασικές εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα, είδαμε διευρύνσεις που έλαβαν χώρα. Τη διεύρυνση τη βλέπουμε θετικά και το κόστος της λήψης αποφάσεων είναι υψηλό όμως. Και αυτό οδηγεί σε αντιδράσει του εκλογικού σώματος και αργούν οι αποφασίσεις, διότι χρειαζόμαστε συνένεση 28 κρατών. Δεύτερον, αντιμετωπίζουμε διάφορες κρίσεις στην Ευρώπη που αθρίζονται και χρειάζονται κατεπίγουσες αποφάσεις από θεσμικά όργανα. Ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα όχι μόνο να λαμβάνουμε αποφάσεις αλλά να τις εφαρμόζουμε επιχειρησιακά. Και για την Προεδρία υπάρχει ιδιαίτερος ρόλος και για τη λήψη αποφάσεων αλλά για την υλοποίηση των αποφασιστέντων. Θα αναφερθώ σε αυτό αργότερα, στη μετανάστευση, όταν θα μιλήσω για τη μετανάστευση. Σε αυτό το πλαίσιο αναφερθήκατε και στην πρόκληση του κράτους δικαίου στην Πολωνία και τη μετανάστευση. Για το κράτος δικαίου είναι σημαντικό, βασικό ζήτημα και αρχή της Ευρωπαϊκής Ανώσεως. Είναι μια από τις αξίες στις οποίες βασιζόμαστε και περνάμε μια εποχή που κινδυνεύουν οι αξίες και πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη σοβαρότατα. Θα το κάνουμε αυτό και σαν Ολλανδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αρχές Φεβρουαρίου θα διοργανώσω μεγάλο σεμινάριο για το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε για το κράτος δικαίου εκτός Ευρώπης έχουμε εύκολα σχόλια. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε και το τι γίνεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το κράτος δικαίου. Θα το θέσουμε το θέμα του κράτους δικαίου και στις δραστηριότητές μας στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Μαΐου για την Πολωνία να πω σε αυτό το στάδιο ότι οι πρόσφατες εξελίξει όσον αφορά το συνταγματικό δικαστήριο και το νόμο δημιουργούν ερωτηματικά για το κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε δύο επιστολέ στην πολωνική κυβέρνηση υπογραμμίζοντας τι κοινέ αξίε, του άρθρου 2, τις κοινέ ευρωπαϊκές Αξίε, είμαι σε επαφή με τον κύριο Γιάνκλαντ, ο οποίο ε, δραστηριοποιείται στον τομέα. Είναι σημαντικό λοιπόν η όλη διαδικασία να προχωρήσει, έχει ήδη ξεκινήσει. Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θεματοφύλακα των συνθήκων ε, υπέχει πρώτη ευθύνη, αλλά βέβαια και το Συμβούλιο ε, υποστηρίζει τη συζήτηση για το κράτο δικαίου. Θα πρέπει να κινηθούμε σεβόμενοι ένα τον άλλον πλήρω, αποκλιμακώνοντας τη ρητορική και να μιλάμε για τα διάφορα ζητήματα μέσω διαλόγου που θα είναι σοβαρός για τη μετανάστευση όπως ανέφερα, όταν μιλάμε για το κάτω δικαίου, η μετανάστευση προβάλλεται και αυτό είναι κάτι που συζητούμε και θα συζητηθεί στο σεμινάριο που διοργανώνουμε. Σε αυτό το πλαίσιο και εσείς και οι συνάδελφοί σας ρωτήσατε ποια η στάση μας για τα μεταναστευτικά, η ύψιστη προτεραιότητα για τις προσπάσεις που καταβάλουμε και ο Ούγγρος συνάδελφος αναφέρθηκε σε αυτό, είναι κρίσιμο ζήτημα. Πρώτα απ' όλα Έχουμε κάποιες αποφάσεις που ελήφθησαν η δράση για την Τουρκία για τη συνέχεια που θα δοθεί στην ε, Βαλέτα, την αναθεώρηση του Δουβλίνου με εγκατάσταση εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεω και πρόταση για μεθοριοφύλακες. Δεν υπάρχει έλλειψη ε, προτάσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέβαλε πάρα πολλέ προσπάθειε τον Δεκέμβριο. Αν δείτε το συνδυασμό των μέτρων θα δείτε ότι είναι λογικά. Κινούνται βάσει τεσσάρων αξώνων και αποτελούν προϋπόθεση για τη λειτουργία των διαφόρων στοιχείων μεταξύ τους. Μετά έχουμε εταιρικέ σχέσεις με τις χώρες, ε, όπως την Αφρική, ε, η Ορδανία, Λίβανο, θέλουμε να προχωρήσουμε εκεί και με την Τουρκία και είπα ύπατη εκπρόσωπος δραστηριοποιείται στην όλη διαδικασία όσον αφορά τη Συρία. Περιπλοκότατο, δυσχερέστατο, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Χρειάζεται προσοχή των πάντων και όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά, η πρόταση για τους μεθοριοφύλακες είναι σημαντικό θέμα, ελπίζουμε να προωθηθεί και θα συζητήσουμε το θέμα της κυριαρχίας και της αποτελεσματικότητας των εξωτερικών συνόρων. Είναι κρίσιμο τομέα προσυζήτηση στο Συμβούλιο και προφανώς και με εσά. Για το θέμα του Σέγγεν και του Δουβλίνου αλληλένδετα, στενά συνδεδεμένα η Ολλανδική Προεδρία ανέλαβε την πρωτοβουλία να εξασφαλίσει, όχι γιατί μας αρέσουν τα τέρμονα συμβούλια, αλλά επειδή υπάρχει τέτοιο θέμα, αναλάβουμε την πρωτοβουλία και τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε ε, μηνιαία μηνιαίες συναντήσεις του Συμβουλίου Εσωτερικών και Δικαιοσύνης ώστε όλα αυτά τα θέματα να προχωρήσουν διότι βλέπουμε ότι τα, οι αριθμοί είναι υψηλοί τα αναφέρατε την εισρωή από απ' έξω από την Ευρώπη και γι' αυτό υπάρχουν κάποιες προτάσεις. Ε, πρέπει να δούμε πώς εφαρμόζονται και ποια είναι η ισορροπία μεταξύ των εφόρων παραγόντων, συμπραγμανών των συζητήσεων που διεξάγονται στην Τουρκία. Όλα αυτά πρέπει να ταιριάξουν, χρειάζεται πάση στηριότητα από όλου μα. Ναι, θέλουμε νομοθεσία, ναι, θέλουμε τα ρυθμίσει, ναι, θέλουμε άνοιγμα, ναι, θέλουμε να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και η Προεδρία σίγουρα θα επενδύσει σε αυτό το τομέα. Οπότε είχαμε σε κάτι άλλο που εφήγει διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο το Δεκέμβριο για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε πραγματικά, συζήτησαν οι ηγέτες το θέμα αυτό που θεωρώ ότι είναι δύσκολο να λυθεί αλλά όχι ανέφικτο. Στόχος είναι να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι όλοι πιστεύουμε ότι είναι καλό για όλους. Στόχος να καταλήξουμε σε κάποια απόφαση στην επόμενη συνεδρίαση το Φεβρουάριο, να δούμε αν τελικά θα το πετύχουμε, δεν δίνω κάποια εγγύηση θα συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τούσκ που έχει πρωτίστως την ευθύνη για να προχωρήσει το θέμα. Μετά από αυτό θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Βρετανικό λαό αν θέλει να παραμείνει ή όχι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Νομίζω ότι ξέρετε τα διάφορα χαρτοφυλάκια είναι πάρα πολύ σημαντικά και όσον αφορά τις νομοθετικές πτυχές, αν κάτι τέτοιο ισχύσει, θα ε, ε, επανέλθουμε σε συζητήση με το Κοινοβούλιο. Κατανοώ πλήρως το θέμα. Το έθεσα. Το λέω ταπεινά, το, το θέμα του εκλογικού νόμου, διότι ε, γνωρίζουμε τις συζητήσεις που διεξάγονται στο Κοινοβούλιο και στη χώρα σας. Και στο Συμβούλιο είναι γνωστή η πρόταση. Και το κείμενο του ΕΛ και τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Εκλογικού Νόμου, κατά την άποψή μου, εμπνέεται τουλάχιστον από κοινή φιλοδοξία, ούτω ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον των πολιτών τη ευρωεκλογία. Ανέφερα κάποια στοιχεία που σε κάποιε χώρε είναι αρκετά χαμηλά, θα πρέπει να το επεξεργαστούμε το θέμα. Επίση, με μεγάλο ενδιαφέρον διαβάζουμε τι προτάσει που υποβάλλατε. Νομίζω την 11η Νοεμβρίου θετήσατε την έκθεση όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου. Εξέτασα όλα τα στοιχεία αυτού, ευρύ φάσμα των προτάσεων Υποχρεωτικό όριο είναι ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού και άλλα στοιχεία περιέχονται στην πρόταση κοινή προθεσμία για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να προτείνουν τους βασικούς υποψηφίους και η ορατότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, ψηφοφορία μέσω διαδικτύου, εναρμονισμένες προθεσμίες. Προφανώς αυτό απαιτεί πάρα πολλές εθνικές κυρώσεις επίσης, επικυρώσεις μάλλον. Ε, είναι ρεαλιστικό να το πούμε. Δηλαδή ότι οι διάφορε απόψει εντό του Συμβουλίου και εντό των διαφόρων κοινοβουλίων υπάρχουν και εντό του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό δεν δίνει μεγάλα περιθώρια λιγμών στο Συμβούλιο, διαφορέ απόψεων δηλαδή. Έχουμε προγραμματίσει προκαταρτική εξέταση του κειμένου σα από το αρμό, φορεί του του Συμβουλίου, 29 Ιανουαρίου θα γίνει. Θα σας ενημερώνουμε για την πρόοδο που ελπίζουμε να υπάρξει ε, για αυτό το θέμα που είναι και ευαίσθητο. Αφορά πολλά πολιτικά κόμματα, πολλά κοινοβούλια και εδώ και στα κράτη-μέλη. Έχουν συγκεκριμένες απο, ε, απόψεις και υπάρχουν διαφορές μεταξύ χωρών. θέλουμε να προχωρήσουμε θα πρέπει να επενδύσουμε πολύ σε προσπάθειες όσον αφορά το μητρό διαφάνειας ο πρόεδρος Γιούνκερ, όπως γνωρίζετε, συμπεριέλαβε την επεξεργασία υποχρεωτικού μητρώου στις πολιτικές του προτεραιότητες και στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εν πάση περιπτώσει ως Προεδρία το βλέπουμε αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για υποχρεωτικό μητρώο το επόμενο εξάμεινο. Τότε βεβαίως θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις επ' αυτού ώστε να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό θέμα για όλους μας να υπάρχει διαφάνεια. Ανέφερα κάποιες από τις δικές μας ιδέες για να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Όσον αφορά το δικαίωμα εξέτασης, ε, βλέπω ότι έχετε μεγάλη αγωνία για το θέμα και απογοήτευση, μεγάλο έργο. Ε, εγώ είμαι από καλβενιστική χώρα και το αίσθημα της ενοχής αρχίζει να με κατακυριεύει. Ε, κοιτάξτε, παντού αν είναι κανείς σοβαρό κοινοβούλιο το δικαίωμα εξέτασης είναι σημαντικό χαρακτηριστικό της εποπτείας και αυτό ισχύει και για σας. Δεν σας αποκρύπτω, το ξέρετε καλύτερα από μένα άλλωστε ότι είναι περιπλοκότατο το θέμα διότι αφορά πάρα πολλά ζητήματα διαφορετικά, τα εξέτασα και στο Συμβούλιο δημιουργούνται προβλήματα θέματα εμπιστευτικότητας, ε, κυρώσει, ε, θέματα μαρτύρων, και υπαλλήλων της, ε, των κρατών μελών. Καλωσορίζουμε τη δέσμευση του εισηγητού να λάβει υπόψη κάποιες από αυτές τις ανησυχίες του Συμβουλίου. Αυτές οι ανησυχίες θα πρέπει να εξεταστούν ομού από κοινού για να λάβουμε, να γίνουν σοβαρές πολιτικές διαπραγματεύσεις. Είναι σημαντικό και προσβλέπουμε σε αυτό να ακούσουμε πώς θα αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του, κοινο... του Συμβουλίου το Κοινοβούλιο. Υπάρχει ένας τρόπος να γεφυρωθεί το πρόβλημα, το αναφέρατε, δηλαδή να υπάρξει τεχνικής φύσεως συνεδρίαση με τον εισηγητή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό ήθελα να πω περί αυτού σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το στάδιο Νομίζω ότι εκάλυψα τις τεθήσεις ερωτήσεις. Ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Ρίτσαρτ, έχεις τον λόγο. Ε, και εγώ σας ευχαριστώ. Για την παρουσίαση που μας κάνατε και για τις προθέσεις που παρουσιάσατε, τις οποίες οπωσδήποτε καλωσορίζουμε. Αναμένουμε τη συνεργασία μαζί σας, αν και όπως είπατε ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Να θέσω ένα άλλο ζήτημα. το Εθνικό σας Κοινοβούλιο είναι ένα από τα πολλά κοινοβούλια που προωθούν την ιδέα της πράσινης κάρτας, όχι κόκκινης, πράσινης, για να προωθούν ιδέες για ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στη χώρα μου αυτό το έχει κάνει η Βουλή των Λόρδων, ε, γιατί στη Βουλή των Λόρδων η πλειοψηφία είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουν να προτείνουν κάτι πιο επικοδομητικό από την κόκκινη κάρτα τη οργανικής κυβέρνηση, οπότε υποστηρίζουν την πράσινη κάρτα. Αυτή τη στιγμή, όπω ξέρετε, σύμφωνα με την συνθήκη, η Κομισιόν έχει το δικαίωμα τη πρωτοβουλία ε, το αποκλειστικό δικαίωμα, δηλαδή έχει αποκλειστικότητα στι ιδέε. Το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από την Κομισιόν να συντάξει μια πρόταση και το Κοινοβούλιο και η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Το σκεπτικό λοιπόν είναι να υπάρξει μια τέταρτη δυνατότητα για να μπορούν π.χ. το 1 τρίτο των Εθνικών Κοινοβουλίων να προτείνουν κάτι τέτοιο στην Κομισιόν. Το έχετε σκεφτεί καθόλου, το έχετε συζητήσει στο Συμβούλιο, γνωρίζω πως ε, ίσως ε, πρώτα θα πρέπει να τοποθετηθεί η Κομισιόν αλλά θα ήθελα να ακούσω τις σκέψεις σας και για να γίνω και λίγο προκλητικός θα μπορούσε κανείς να πει πως ε, το αίτημα αυτό επιδεικνύει και αποδεικνύει πως τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν εμπιστεύονται το Συμβούλιο Αλλιώς ε, δεν θα υπήρχε ανάγκη για κόκκινη, πράσινη ή μπλε ή οτιδήποτε άλλη κάρτα. Υποτίθεται ότι οι κυβερνήσει σέβονται τα εθνικά κοινοβούλια. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ε, το έχετε συζητήσει καθόλου στο Συμβούλιο αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ κύριε Τάνεμαντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Κούντερς. Είμαι μέλος της ομάδας ε, ENF, συνεργαζόμαστε με τον κύριο Βίλντερς, ο οποίος εδώ πέρα είναι αντιπολίτευση βεβαίως και ε, δεν είναι όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια ομοσπονδιακή λογική, ούτε θεωρούμε πως είναι πάντα η καλύτερη λύση. Και δεν είναι ανάγκη να μιλάτε με, θρησκευτικά, με θρησκευτική ρητορία και όταν δεν πιστεύουμε στην Ευρώπη να μας λέτε ότι ε, είμαστε εγωιστές και εθνικιστές όπως κάνει και ο κύριος Λάινεν. Απλά μπορούμε να αμφιβάλλουμε και να αμφισβητούμε το εάν το κάθε πρόβλημα μπορεί να λυθεί με μια κοινοτική λύση. Αυτό κάνουμε. γιατί συνεχώς πηγαίνουμε προς ε, την ομοσπονδιακή σκέψη και συνεχώς ζητάμε περισσότερη ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα σε αυτή την Επιτροπή που έχουμε διάφορα σχέδια ε, ε, εντός ε, της ε, συνθήκης Λισαβόνας αλλά εδώ πέρα και ο κύριος Φερχόστατ μας είπε πως ό,τι δεν μπορεί να γίνει εντός της συνθήκης θα απαιτήσει μια αλλαγή αυτής. Είπατε πως λοιπόν πάρα πολλοί αναζητούν λύσεις και στρέφονται προς την Ευρώπη αλλά ξέρετε και αυτήν Ολλανδική εμπειρία πως ε, δεν συμβαίνει πάντα αυτό ή δεν ε, μπορεί να συμβαίνει πάντα. Λοιπόν, η ερώτησή μου κάπως ρητορική είναι, θα τα λάβετε υπόψη καθόλου όλα αυτά. Η Μάιτε Ρουίς, ευχαριστώ και καλώς ήρθατε κύριε Κούντερ, κύριε Υπουργέ. Η αλήθεια είναι ότι επιθυμούμε διακαώς να στεφθεί με επιτυχία το εξάμεινο της Ολλανδικής Προεδρίας. Γιατί σίγουρα το 2015 δεν θα περάσει στην ιστορία ως ε, η καλύτερη χρονιά από την άψη της συμβολής του Ευρωπαϊκού του Συμβουλίου. Και εσείς είπατε ότι θέλετε να σημειώσουμε πρόοδο σε θέματα διαφάνειας και άλλα θέματα που μπορεί να μην είναι τα πιο κατεπήγοντα, δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αλλά που σίγουρα αφορούν κέρια ζητήματα. Γιατί σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα ουσιαστικά αφορούν την ομοποίηση και την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Πέραν τη διαφάνεια και είμαι βέβαιο ότι όλο ο κατάλογο των θεμάτων που μα αναφέρατε και που αναφέρουν το, την καλύτερη νομοθεσία, καλό θα ήταν να αναπτυχθούν με ενέργεια και ενθουσιασμό όπω υποσχεθήκατε. Πέραν τη διαφάνεια όμω, θέλουμε συνεπή αποτελέσματα γιατί μεταξύ αυτών των συμφωνηθέντων στο Συμβούλιο το 2015 για τα σοβαρότερα θέματα της προσφυγικής κρίσης ε, των συνόρων, μεταξύ των συμφωνηθέντων και των ε, μέτρων που εφαρμόστηκαν, υπάρχει ε, μια άβυσος ασυναρτησίας και έλλειψη συνοχής. Το 2015 λοιπόν ήταν σχετικά άδοξο. Ελπίζουμε το 2016 να είναι διαφορετικό, να περάσει στην ιστορία σημαντική χρονιά και να κάνετε εσεί την αλλαγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κρίση μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας, που έχει τεράστια σημασία ε, σε ό,τι αφορά τις διπλωματικές ε, απόπειρες αναζήτησης ε, λύσης σε όλα τα θέματα που άπτονται της παγκόσμιας τρομοκρατίας, του συριακού προβλήματος. Έχετε καμία ελπίδα να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και να βρεθεί μια λύση. Βραχυπρόθεσμα, ευχαριστώ και καλή σας τύχη. Ευχαριστώ Μαϊτή και να ολοκληρώσω με τα δικά μου σχόλια. Το γύρο αυτό αναφερθήκατε στην Διοργανική Συμφωνία για την Καλύτερη Νομοθεσία που αποτελεί και πρόκληση και της δικής σας Προεδρίας. Στο Κοινοβούλιο πόρο απέχουμε, δεν ξέρω πόσο, αλλά πόρο απέχουμε από την έγκριση στην Ολομέλεια ώστε ο Πρόεδρος μας να υπογράψει με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Συμφωνία. Και μάλιστα θα έχουμε και νέα έκθεση για την εφαρμογή, δηλαδή για την ερμηνεία της διοργανικής συμφωνίας και τους μηχανισμούς εφαρμογής. Εκεί μερικά θέματα αφορούν τις εσωτερικές μας δομές και τις πιθανές αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν σε... στο καταστατικό μας, στον ιστορικό μας κανονισμό. Πάντως κάποιες πτυχές ε, θα πετήσουν στενότερη συνεργασία μεταξύ των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και ευελπιστώ μια και ασχοληθείτε με τα θέματα της εφαρμογής ε, ε, ίσως χρειαστεί να ξανακαθίσουμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων με Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσβλέπουμε σε αυτό στη δική σας προσέγγιση και στην ε, δική σας καλή βούληση ώστε να γίνει πιο θελκτική αυτή η συμφωνία που δεν εκ πρώτης τόσο ελκυστική και τα θέματα της δημοκρατίας, της αποτελεσματικότητας, ε, της νομοποίησης ε, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και τους πολίτες. Οπότε μια αίσια έκβαση θα χαιρετηθεί πιστεύω από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτά τα σχολεία μας. Ε, έχετε και πάλι το λόγο κύριε Υπουργέ. Thank you very much, Madam. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και τις ερωτήσεις των συναδέλφων για τη σχέση μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων και εθνικών κοινοβουλίων και της ευρωπαϊκής θέσπισης πολιτικής. Τα εθνικά κοινοβούλια πραγματικά πιστεύω, βλέποντας τη χώρα μου, θεωρώ ότι έχουν μηχανισμό τεράστιο για να ελέγχουν τις εθνικές κυβερνήσεις πώς τοποθετούνται αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα εθνικά κοινοβούλια είναι τα μόνα θεσμικά όργανα. Έχουμε δημοψήφισματα και πρωτοβουλίες πολιτών ούτως ώστε αντικατοπτρίζονται οι πράξεις των, εθ... οι πράξεις των εθνικών κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλουμε να στηρίζεται από τον πληθυσμό και τα καταφέρνουμε πάντα το ότι τα εθνικά κοινοβούλια θέλουν να είναι πιο δραστήρια στη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρώ ότι είναι αρνητικό, αντίθετα το κατανοώ. Ε, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξελιχθεί, έχει βρει έναν τρόπο ε, να διοργανώνεται κατά ανάγκη, συμμεριζόμαστε την κυριαρχία και τα εθνικά κοινοβούλια θέλουν να παίξουν ρόλο. Αυτό δεν εκφράζει απαραίτητα έλλειψη εμπιστοσύνης ε, έναντι εθνικών κυβερνήσεων. Βλέπω ότι ενδιαφέρονται να συζητούν μαζί σας, να συζητούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελέγχοντας τα όσα πράττουν οι κυβερνήσεις μας στις Βρυξέλλες και αυτό καθ' αυτό θα πρέπει να βοηθήσει. Τώρα για τις ε, πράσινες κάρτες, η εισαγωγή κυτρίνων και πρασίνων καρτών θα ε, σήμαινε μια αλλαγή ε, των ε, διαφόρων πρωτοκόλων των συνθήκων. Κυρίως αν θεσπιστεί μια διαδικασία επίσημη πράσινης κάρτας, αυτό επιτυχάνεται μόνο μέσω αλλαγής συνθήκων και αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω των ισχυουσών συνθήκων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πολλά να αυξήσει τι επαφέ μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπογραμμίζουμε την σημασία που έχουν στενέ επαφέ αυτέ. Πάνω από 200 φορές υπήρξαν επισκέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Εθνικά Κοινοβούλια. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία των στενών επαφών μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικών Κοινοβουλίων στον αφορά την πρωτοβουλία για τη δικασία της πράσινης κάρτας. Πώς θα λειτουργούσε αυτό. Κάποιοι είπατε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Προφανώς πρέπει να υπάρχει μια συνεπής άποψη όσον αφορά ε, τις αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό στο πλαίσιο αυτό τα εθνικά κοινοβούλια να λάβουν τα ίδια πρωτοβουλία όπως το κάνουν στη χώρα σας, στη δική μου και σε κάποιες άλλες. Ε, οι συζητήσεις ξεκίνησαν ήδη στην Κόσακ μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων όπως συνεδρίασε της Κόσακ στις 30 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο. Είναι ένα βήμα για αλλαγέ αν θέλετε. Το Συμβούλιο υποστηρίζει την εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διαδικασία Ευρωπαϊκή Διαμόρφωση Πολιτικών Γι' αυτό το λόγο γίνονται αναφορέ στο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στη Γερμανική Συμφωνία για καλύτερη θέσπιση νομοθεσιών και η, η εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων αυξάνει την ευρωπαϊκή νομιμότητα. Να δούμε πώς θα γίνει, πώς θα ληφθεί αυτό υπόψη διαπραγματεύσεων του Ρωμένο Βασίλειο και πώς αυτό θα οδηγήσει σε προτάσεις ή όχι. Εν πάση περιπτώσει αυτά είχα να πω σε αυτή τη φάση τα εθνικά κοινοβούλια είναι φορείς που θα πρέπει να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες. Ε, όσον αφορά την αντίδραση, την αντίθεση της ενστάσεις και την αντιπολίτευση. Σαν πραγματικός δημοκράτης θεωρώ ότι είναι κρίσιμο να ακούγονται όλες οι φωνές και στο Ευρωκοινοβούλιο όπως γίνεται στα Εθνικά Κοινοβούλια. Νομίζω ότι υπάρχει έντονη συζήτηση όσον αφορά την Ευρώπη ε, στις χώρες μας όλες με διαφορετικές απόψεις ευρωσκεπτικιστές που είναι κατά της Ευρώπης ε, αυτοί που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδιοποίησεως ξέρετε όλες τις απόψεις που υπάρχουν είναι πολύ σημαντικό όλες οι απόψεις να λαμβάνονται υπόψη σοβαρά θα το κάνει αυτό προφανώς το Συμβούλιο θα τις λάβει όλες υπόψη του θα έλεγα από τη δική μας σκοπιά σε αυτή τη φάση βλέποντας τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη ανεξαρτήτως απόψεως είναι σημαντικό για θέματα όπως είναι το άσυλο και η μετανάστευση και η τρομοκρατία να υπάρχει αποτελεσματική ευρωπαϊκή συνεργασία για να αντιμετωπιστούν οι απειλές και τίθεται θέμα εθνικής κυριαρχίας όσον αφορά τις ευρωπαϊκές δράσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει σχετικώς προτάσεις και θα αποφασίσουμε. Και θα συζητηθούν τα θέματα αυτά και εδώ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όσον αφορά Συρία, Ιράν, Σαουδική Αραβία, ίσως να είναι εκτός των θεμάτων αυτής της Επιτροπής, να πω ότι με τις εκτελέσεις στη Σαουδική Αραβία που είπατε εκπρόσωπος και εγώ Υποστηρίζουμε συγκεκριμένη θέση. Θεωρούμε ότι παραβιάστηκε το κάτω δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα και σοβαρότατα δημιουργήθηκαν μεγάλε εντάσεις με το Ιράν που και εκεί υπάρχει η θανατική ποινή και υπάρχει και αντιπαλότητα γεωπολιτική μεταξύ των δύο χωρών και έχει, ε, έχουμε πάρα πολλούς πολέμους αντιπροσώπων που γίνονται στην περιοχή όπως και στη Συρία. Διπλωματικές προσπάθειες όλων κατευθύνονται μέσω της ΥΠΑ του Στην αποκλιμάκωση των εντάσεων. Υπάρχει διπλωματική συμφωνία με το Ιράν. Αρνητικά τα αποτελέσματα. Αυτά που συνέβησαν μάλλον είναι αρνητικά. Ο κ. Ντεμιστούρα συναντήθηκε, ο ειδικό εκπρόσωπο για τη Συρία, με του αρμοδίου. Να εξεταστεί κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της διαπραγματεύσης στη Γενέβη και στη Νέα Υόρκη για τη Συρία. 25 Ιανουαρίου έχει πραγματιστεί η συναντρίαση και οι δύο πλευρές είπαν ότι θα συμμετάσχουν. Παραδόξως, η ύπαρξη διαπραγματεύσεων μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση και σε προσπάθειες συνεργασία για να καταπολεμηθούν οι φρικαλαιότητε που βλέπουμε στη Συρία και να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης για ανθρωπιστική βοήθεια. Κυρία Πρόεδρε, ρωτήσατε κάποια πράγματα. Απατώντας λέγω ότι πρέπει να συνεργαστούμε επικοδομητικά για ταχύ εφαρμογή της συμφωνίας ούτω ώστε να εφαρμοστεί στην δεύτερη θητεία, στο δεύτερο ήμιση τη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καθήκον όλων των θεσμικών φορέων. Θα συνεργαστούμε στενά για να εφαρμοστούν στις διατάξεις για τη διαφάνεια θα πρέπει να ξεκινήσουμε να βελτιώσουμε το θέμα της ανιχνευσιμότητας της νομοθετικής διαδικασίας, η βάση δεδομένων να είναι φιλική προς το χρήστη, συμφωνία για αμοιβή ανταλλαγή απόψεων, τριμερείς διαλόγους κλπ. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όσον αφορά τις απόψεις μας. Το βλέπω ευνοϊκά το θέμα, βλέπω ευνοϊκά τη συνεργασία μας Συγχαίρουμε προφανώς τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία που επιτυχώς ολοκλήρωσε τις προσπάθειες, τη Διοργανική Συμφωνία για καλύτερες ρυθμίσεις, καλύτερη νομοθεσία. Ελπίζω η επίσημη επισήμως να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας το ταχύτερο δυνατόν και μετά βέβαια να υλοποιηθούν τα αποφασιστέντα που αυτό είναι το σημαντικότερο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω εδώ ολοκληρώνουμε τη συνεδρίασή μας με την, τη συνάντησή μας με την Προεδρία. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κάτι κατεπήγον για να αγκαστούμε να σας προσκαλέσουμε σύντομα. Ε, ελπίζουμε ότι στο τέλος τελικά θα έχετε κάτι να μας πείτε, θα έχετε να παρουσιάσετε επιτυχής προεδρίας, ε, προσευχόμεθα γι' αυτό και θα βασιστείτε και στην συνεργασία μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ολοκληρωθήκε η συνεδρίαση, παρακαλώ να μην τις θέσεις. Έχω σημαντικά πράγματα να σας πω. Uh, Συνάδελφοι, θέλω να εκμεταλλευτώ κάθε λεπτό του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας. Μια στιγμή γιατί έλαβα ένα αίτημα του κυρίου Γιασδόφσκι, που είναι εισηγητής της έκθεσης για την ετήσια έκθεση του 2014 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα πιέζεται λόγω των, ε, του φορτωμένου προγράμματος που έχει ε, και μου ζήτησε να διεκπαιρεώσουμε το συντομότερο δυνατό την έκθεση. Δεν είναι προβληματική, δεν υπάρχει διάσταση απόψεων, οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να την διεκπαιρεώσουμε τώρα στο τέταρτο που μας έχει απομείνει για να τελειώσουμε νωρίτερα το απόγευμα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γιασδόφσκι για να μας παρουσιάσει την ε, έκθεσή του. Θα μιλήσω πολωνικά. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για μια συμπληρωματική έκθεση που συμπληρώνει την έκθεση Επιτροπής ε, ε, Νομικών Υποθέσεων που είναι κατ' ουσία αρμόδια για το θέμα αυτό. Εμείς στη γνωμοδότηση ε, εκδίδουμε και είναι απόδειξη μια συνέχεια των εργασιών μας γιατί θα θυμάστε τη γνωμοδότηση του 2013 για την εφαρμογή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας ε, για το 2013 ε, που εγκρίναμε σχετικά πρόσφατα πριν από μερικούς μήνες. Στην γνωμοδότηση εκείνη την προηγούμενη προσπάθησα να ασκήσω πίεση ε, ως προς την ανάγκη εφαρμογής των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και αυτό αφενός αναφέρεται στην, στον όλο και μικρότερο αριθμό αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά έχουμε και σημαντικές συστάσεις. Προτείνω πολύ σημαντικές συστάσεις, όπως είναι η έντονη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε ο διάλογος και μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικών Κοινοβουλίων ε, να γίνει όλο και πιο εντατικός. Προτείνουμε, όπως και στην προηγούμενη γνωμοδότηση, ελαστικότερη αντιμετώπιση της προθεσμίας των 8 εβδομάδων που δεσμεύει τα Εθνικά Κοινοβούλια και επίσης ε, έχουμε και μια άλλη ιδέα που την ε, επαναλαμβάνουμε από την προηγούμενη γνωμοδότηση και την ανέφερε προηγουμένως στη συζήτηση με τον Υπουργό και κύριο Κόρμπετ είναι αυτή η σκέψη της ε, πράσινης ε, κάρτας ε, προκειμένου να αποτελέσει την έκθεση ανάμεξης ενεργοποίησης των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και ως έκφραση σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας. Η γνωμοδότησή μου, όπως σας είπα, είναι συμπληρωματική σε σχέση με τις εργασίες της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων που είναι και η καθήλη αρμόδια. Εγώ επικεντρώνομαι στην έκφραση υποστήριξης προς τα Εθνικά Κοινοβούλια ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος του στην προσπάθεια εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας θέλουμε πιο δραστήριο ρόλο και των Εθνικών Κοινοβουλίων εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιο τον λόγο. Λοιπόν, προθεσμία για τροπολογίες προτείνω να μην είναι πολύ μεγάλη. 21 Ιανουαρίου, 6 το απόγευμα. Και ελπίζω όλοι οι συνάδελφοι να προλάβουν. Μια εβδομάδα ολόκληρη. 21 πρώτου, 6 το απόγευμα. Ελπίζουμε να ψηφιστεί στις 14-15 Μαρτίου. την επόμενη συνεδρίασή μας και μετά τα υπόλοιπα εξαρτώνται από την κατά κύριο λόγο αρμοδία επιτροπή. Α, με συγχωρείτε. Μπερδεύτηκα. Ο κύριος Πρέντα, σκιώδης ηγητής του ΕΛΚ, απουσιάζει. Μου έχει αφήσει ένα γραπτό σημείωμα, να σας το διαβάσω. Ευχαριστεί τον κύριο Βιαζόφσκι, θεωρεί πως είναι σημαντικό να συζητηθούν αυτά τα ζητήματα. Λυπάται όμως για το ότι δεν αναφέρεται το ζήτημα της επικορικότητας και νολογικότητας πιο θετικά Μάλιστα η έκθεση του 2014 λέει πως η αρχή της επικουρικότητας και αναλογικότητας έγινε σεβαστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός πως δεν υπήρχε διαδικασία κίτρινης κάρτας δεν σημαίνει πως ε, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την αρχή της επικουρικότητας. Ε, απλά η αρχή δεν παραβιάστηκε. Το νέο πακέτο καλύτερης νομοθεσίας είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, θα ήθελα να πει πως οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να δουν το ζήτημα θετικά, να ενθαρρύνουν τη συζήτηση με τα εθνικά κοινοβούλια, ειδικά στο πλαίσιο του Brexit. Αν τα εθνικά κοινοβούλια δεν θεωρούν ότι συμπεριλαμβάνονται αρκετά, πρέπει να επικοινωνήσουμε καλύτερα για τα μέσα που έχουν στην διάθεσή τους, για να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Νομοθετική Διαδικασία. Οι διακοινοβουλευτικές συναντήσεις είναι πολύ χρήσιμες, πρέπει να τις χρησιμοποιούμε καλύτερα και δεν θα πρέπει τα Εθνικά Κοινοβούλια να θεωρούμε ότι μπλοκάρουν μόνο την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία κατόπιν. Πιστεύει πως δεν χρειάζεται νέος μηχανισμός, γιατί έχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα στη διάθεσή μας για να ελέγχουμε την επικουρικότητα και την αναλογικότητα όπως αναφέρουν οι συνθήκες και πρέπει να μην διακυβευθούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών, ειδικά το αποκλειστικό δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας της Κομισιόν. Αυτά από τον κύριο Πρέντα. Και ο εισηγητή του ΕΛΚ. Τώρα λοιπόν μπορούμε να ολοκληρώσουμε. 21 πρώτου ή προθεσμία για σε έξω το απόγευμα και σας ευχαριστώ κύριε Βιαζόφσκι και ας ελπίσουμε να ολοκληρώσουμε εγκαίρως τώρα να σας πω πως λύεται η συνεδρία διακόπτεται η συνεδρίαση με συγχωρείτε για τις 3 το απόγευμα